So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen, natürlich auch die Dolmetscher. Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Να σας καλωσορίσω, να καλωσορίσω και τους διερμηνείς αλλά και τους επισκέπτες μας σήμερα το πρωί. Έχουμε μία αλλαγή στην ημερήσια διάταξη. Η ψηφοφορία στο σημείο 25 που είναι ε, σχετικό με τον κανονισμό του 2005 θα αναβληθεί. Ε, δεν ξέρω αν υπάρχουν παρατηρήσεις για την ημερησία. Εάν όχι, εγκρίνεται με αυτήν την αλλαγή. Ε, μου φαίνεται ότι όλοι συμφωνούμε, οπότε εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Έγκριση των πρακτικών ε, του Οκτωβρίου 2018. Επίσης, εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, είναι να εγκρίνουμε τη ε, πρακτικά της συνεδρίασης του Οκτωβρίου 2018. Δεν υπάρχουν αντιρρήσει. Σημείο 3. Ανακοινώσει του Προέδρου. Καμία ανακοίνωση δεν έχω εγώ από πλευρά μου, οπότε μπορούμε να μπούμε στην ουσία της ε, ημερήσιάς μας διάταξης, δηλαδή σημείο 4 αυτόνομη οδήγηση στις ευρωπαϊκές μεταφορές. Εισηγητής είναι ο κύριος Φαντεκάμπ, στον οποίο και δίνω άμεσα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ολοκληρώσαμε μία εξαιρετικά θετική και επικοδομητική διαδικασία για την κατάρτιση αυτής της έκθεσης και, με την, ε, και χάρη μάλλον ε, και στην στήριξη της γραμματείας ΕΤΡΑΝ που πάντα ε, μας βοηθά ιδιαίτερα στην διατύπωση των συμβιβαστικών τροπολογιών. Εξετάσαμε διάφορες πτυχές της αυτόνομης οδήγησης ή των αυτόνομων οχημάτων. Δεν πρέπει δηλαδή μόνο για αυτοκίνητα και φορτηγά, αλλά και για το σιδηροδρομικό τομέα και για το μετρό και για σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοείας αλλά και για τα drones, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη τα αναφέρουμε ακροθυγώς. Η έκθεση ιδίω πρωτοβουλία είναι σημαντική γιατί πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει θέση ε, σε σχέση και με τον ανταγωνισμό της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ευρώπη έχει επαρκές ε, δυναμικό και κεφάλαιο ε, για να σημειώσει πρόοδο, όμως ε, δεν πάει αρκετά γρήγορα η διαβούλευση μεταξύ Κομισιών, Κοινοβουλίου και 28 κρατών μελών. Πρέπει λοιπόν να σημειώσουμε πρόοδο σε αυτό το τμήμα. Επισημάναμε και τις κοινωνικές διαστάσεις του φακέλου. Πολλοί πολίτες ακόμα δεν εμπιστεύονται τα αυτόνομα οχήματα και μάλιστα ο κύριος Βαν ε, Μίλτενμπουργκ ανέφερε ότι θα πρέπει να κάνουμε και κάποιες μικρές τροποποιήσεις ε, στο σύστημα κατάρτισης γιατί θα μπορούσαν να υπάρξουν επιπτώσεις εκεί. Σύστημα εκπαίδευση και κατάρτιση. Ε, υπάρχουν ακόμα δύο βασικέ διαφορέ μεταξύ τη πλειοψηφία του κοινοβούλου, από ό,τι φαίνεται, και εμού. Αυτό αφορά την παροχή δεδομένων μέσω των ε, παρασκευαστών, των κατασκευαστών μάλλον. σε σχέση και με τις ε, υπηρεσίες που παρέχονται μετά την πώληση γύρω από ε, τα αυτόνομα Μετά έχουμε και τις, ε, τον κλάδο του leasing που θέλει να έχει όλα τα δεδομένα για τα προγράμματα συντήρησης των αυτοκινήτων αλλά έχουμε και τη διασύνδεση με ξενοδοχεία, με εστιατόρια, αλλά και με το σπίτι μας στο μέλλον. Είναι το γνωστό που μας λένε ότι θα μπορούμε να βάζουμε τη θέρμανση, να λάβουμε τη θέρμανση στο σπίτι μας από τα μάξι πριν φτάσουμε εκεί. Μετά υπάρχουν και άλλα κάποια σημεία ε, σε ό,τι αφορά το λεγόμενο extended vehicle και έτσι συλλέγονται δεδομένα από τους κατασκευαστές και μετά διατίθενται ε, στους ε, υπόλοιπους εταίρους. Ή ε, αν θα δώσουμε τέτοια άμεση πρόσβαση σε όλα αυτά τα δεδομένα. Εγώ ξέρετε είμαι από το ΕΛΚ, είμαι μετριοπαθή σε ό,τι αφορά αυτά τα δεδομένα. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει μία ισορροπία μεταξύ των OAMs και των υπολείπων εταίρων. Όμως άλλοι συνάδελφοι θέλουν να υπάρχει αυτή η άμεση πρόσβαση. Αύριο θα αποφασιστούν όλα αυτά στην ψηφοφορία, εκτός κι αν έρθει κάποιο ευφυή e e συνάδελφο με μια καταπληκτική συμβαστική πρόταση. Αλλά προ το παρόν δεν έχει φανεί κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ και πάλι για τη διαδικασία. Ακούσαμε πολύ καλά λόγια και για την ποιότητα ε, της ε, γνωμοδότησης, της έκθεσης. Υπάρχει βέβαια αυτό το σημείο για τα δεδομένα και ε, στο CITS ε, και στη τη γνωμοδότηση υπήρξε μια διαβούλευση, αλλά δεν τα καταφέραμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σιγητά. Και τώρα θα ακούσουμε τη γνώμη των σοσιαλιστών. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας, συνάδελφοι. Πρέπει να ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματος του συναδέλφου Ουλιεβίτς, που, τον οποίο αντικαθιστώ. Πρώτα απ' όλα είμαι πεπισμένος ότι αυτή η έκθεση αποτελεί μια θετική εξέλιξη και θα γίνει θετικά δεκτή από τις διάφορες επιτροπές ε, της, ε, του, του, του Κοινοβουλίου. Μάλλον έγινε θετικά δεκτή και ευχαριστώ τον εισηγητή για το συντονισμό με όλες τις επιτροπές. Ωστόσο υπάρχουν κάποιες ε, παρατηρήσεις που θα ήθελα να κάνω ε, και αυτά σχετίζονται και με την έκθεση CDS που ψηφίσαμε πριν από λίγες εβδομάδες. Οφείλουμε να αγγίξουμε και τα θέματα απασχόλησης και τα κοινωνικά ζητήματα. Σε κάποιες από τις ε, όντως μιλήσαμε για αυτά τα θέματα, όμως πρέπει να ε, τονίσουμε περισσότερο τα θέματα τα κοινωνικά. Γιατί δεν ζητάμε με πιο ε, άμεσο και ξεκάθαρο τρόπο μια γενική στρατηγική από πλευράς της Κομισιόν. Χρειαζόμαστε περισσότερες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Η αυτοματοποίηση, αυτή η νέα βιομηχανική επανάσταση τρέχει. Δεν έχουμε χρόνο να χάσουμε. Έχουμε φτάσει λοιπόν σε αυτό το σημείο. Παράγραφοι 4 και 4α. Μιλάμε για την ε, ε, ιδιοκτησία των δεδομένων για μια νομική πρόσβα, ε, κάλυψη όσον αφορά την ουδέτερη πρόσβαση, τεχνολογική πρόσβαση στα δεδομένα για ολόκληρη την αλυσίδα αξίας ε, του τομέα των αυτοματοποιημένων οχημάτων. Στην έκθεση για την στρατηγική για τα συνεργατικά ευφύ συστήματα μεταφορών θέλουμε ε, να μιλήσουμε για ολόκληρη την αλυσίδα. Τώρα γίνονται απόπειρε ε, να, περιοριστούν, ε, να περιοριστεί η νομική κάλυψη. Χθε το βράδυ το ΕΛΚΑ και η ΑΛΔΕ έδειξαν τη στάση του απέναντι σε αυτές τις συμβαστικές τροπολογίε. Αφού απορρίφθηκαν διάφορες προτάσεις, ο κύριος ε, Φαντερκάμπα βελτίωσε την ε, θέση, αλλά παραμένουν διαφορές. Χρειάζεται νομοθετική πρωτοβουλία, όχι μόνο στρατηγική από πλευράς της Κομισιόν με την συμμετοχή ολόκληρης της αλυσίδας αξίας και όχι μόνο ε, ένα τμήμα των τρίτων μερών. Αυτή είναι η θέση των σοσιαλιστών και του σκιώδη εισηγητή του κύριου Ουλιεβιτς. Μάλιστα, ευχαριστώ και ευχαριστώ που αντεκαταστήσατε τον συνάδελφο να ακούσουμε το τώρα τον κύριο Σλοτόφσκι από το ECR. Sprawozdawcy, panu Van de Kampowi oraz kolegom sprawozdawcom cieniom za dotychczasową pracę nad tym raportem. Nie chciałbym tutaj powtarzać po raz kolejny tych samych argumentów. Ευχαριστώ τον σκιώδη συγητή. Δεν θα επαναλάβω τα επιχειρήματα που ήδη παρουσιάστηκαν όσον αφορά την ε, αυτόνομη οδήγηση. Εδώ και καιρό ασχολούμαστε με αυτή την έκθεση και οι τροπολογίες μας έχουν να κάνουν ε, με την ασφάλεια και την προστασία των καταναλωτών. Η ομάδα ECR επιθυμεί να ε, υπάρχει θεμητός ανταγωνισμός όσον αφορά τη συντήρηση αυτών των αυτόνομων ε, οχημάτων. Η εισαγωγή αυτόνομων οχημάτων <coughs> θα έχει αντίκτυπο για τα συνεργεία αυτοκινήτων. Η πρόσβαση στα δεδομένα έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Σίγουρα βέβαια πρέπει να υπάρχουν ε, και μέτρα ασφαλεία ε, και προστασία των ε, πνευματικών δικαιωμάτων. Υπάρχει πραγματικά κίνδυνος να υπάρχουν κενά στην ασφάλεια και γι' αυτό θα πρέπει όλα αυτά τα θέματα να λεφθούν πολύ σοβαρά υπόψη ένα μελλοντικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Θεωρούμε ότι άμεσα θα πρέπει να γίνουν τα απαραίτητα νομοθετικά μέτρα. Όχι όμως να ορίσουμε προθεσμίες που είναι μη ρεαλιστικές. Αυτή η προθεσμία το 2020 ε, νομίζω ότι είναι λογική, αλλά κατά τα λοιπά συμφωνώ με τις νέες συμβιβαστικέ προτάσεις και με την έκθεση και η ομάδα μας θα ψηφίσει υπέρ της έκθεσης. Ευχαριστούμε κύριε Σιλωτόφσκι. Θα ήθελα τώρα να παρακαλέσω τον σκιώδη συγκητή από την Άλντε, Φαν Μίλτεμπουργκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Βαντεκάμπ και τους σκιώδης συγητές για μια σημαντική έκθεση γιατί νομίζω ότι μπορούμε έτσι να σημειώσουμε ένα βήμα ακόμα στην προσπάθεια αυτή αυτόνομων οχημάτων ε, στην Ευρώπη. Και σημαντικό είναι να είμαστε και ηγέτιδα δύναμη, γιατί και οι υπόλοιπε περιφέρειε του κόσμου δεν ε, κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια. Ε, σημαντική είναι η συμβολή των αυτονόμων οχημάτων και προ την μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Θεωρώ ότι αυτό σωστά αναφέρεται και στι τροπολογίε και στι συμβαστικέ. Όλε οι τροπολογίε που αφορούν την τεχνικά ουδέτερη προσέγγιση και την δίκαιη πρόσβαση στα δεδομένα. Τα έχουμε συζητήσει ήδη. Σημαντικό είναι να έχουμε εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Υπήρξε μια συζήτηση για την παράγραφο 4 και 4α. Χαίρομαι που οι εισηγητές τώρα έχει αναφέρει και έχει προσθέσει τον όρο νομοθεσία και αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό να εντοπίσουμε ποιε είναι οι απαραίτητε κανονιστικέ ρυθμίσεις. Εγώ μπορώ να δεχτώ τη συμβαστική τροπολογία αυτή τη στιγμή, αλλά φαίνεται ξεκάθαρα ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρχει ρύθμιση, κανονιστικό πλαίσιο. Και νομίζω ότι πρέπει να γίνει αυτό σε ό,τι φορά τα αυτόνομα οχήματα, γιατί δεν είναι μόνο θέμα δημοσίου συμφέροντο. αλλά και για να δώσουμε κίνητρα στην καινοτομία και η πρόσβαση στα δεδομένα είναι σημαντική και από αυτήν την άποψη. Κλείνοντα, Πρόεδρε, είναι σημαντική αυτή η έκθεση και δίνει σημαντικέ κατευθύνσει και προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η νομοθεσία είναι απαραίτητη και με την μνήα που έκανε και ο εισηγητή ότι είναι σημαντικό να εξετάσουμε με μεγάλη προσοχή τι ακριβώ είναι απαραίτητο, να γίνουν αξιολογήσει αντικτύπου. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι δεν χρειάζεται όποιος φτιάχνει ένα όχημα να έχει και πρόσβαση σε όλα τα, όχημα σε όλα τα δεδομένα απαραίτητα. Θα τα δούμε στην πορεία, θα στηρίξουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζουμε να υπάρχει ευρία συνένεση και ευρία πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, γιατί νομίζω ότι έτσι θα αυξηθεί και η σημασία της ε, έκθεσης για την Επιτροπή. Ευχαριστώ και περιμένω την ψηφοφορία. Ευχαριστούμε πολύ κύριε δεν βλέπω άλλους κοιόδης εισηγητές ε, στην αίθουσα τους πρασίνους για την αυτόνομη οδήγηση. Δεν υπάρχει κάποιος που το λόγο. Αν όχι, από την Επιτροπή ΕΟΚΕ, ο εκπρόσωπος παρακαλώ να πάρει το λόγο. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μου δώσετε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω τη δική μας γνωμοδότηση για τη συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα. Εμείς στηρίζουμε την πρωτοβουλία και μάλιστα θερμά, διότι θεωρούμε ότι η τεχνολογία είναι πλέον αρκετά όρημη, ώστε και στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας να φτάσουμε σε πρότυπα ασφαλείας αντίστοιχα με αυτά που βλέπουμε στις αεροδρομικές ή τις αεροπορικές μεταφορές. Ε, για την ε, αυτοματοποιημένη τεχνολογία στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Έχουμε σίγουρα ε, θετικά να πετύχουμε με τις μηδενικές έως εκπομπές, αλλά υπάρχει και πολλή δρόμος μπροστά μας. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει ε, καταρχάς ε, με την ε, υποβοηθούμενη, δηλαδή την ήμι αυτοματοποιημένη οδήγηση και έπειτα θα περάσουμε στην αυτόνομη, διότι υπάρχουν, τελ... υπάρχουν διαφορετικά προβλήματα με μια γρήγορη εισαγωγή. Σε ό,τι αφορά την υποβοήθηση, το σύστημα αυτό, αυτό συνδέεται με πάρα πολλές δαπάνες και μόνο τα καινούργια οχήματα ε, μπορούν να αποφεληθούν αυτή τη τεχνολογία. Δεν γίνεται να εξοπλιστούν αυτή την τεχνολογία τα ήδη κυκλοφορούντα. Ε, και αυτό είναι μεγάλο τροχοπέδι. Έπειτα, ήδη σήμερα υπάρχουν συστήματα υποβοήθησης στα οχήματά μας και όποιοι παρακολουθούν ε, το φαινόμενο αυτό βλέπουν ε, ότι μπορεί κανείς εύκολα να το ακολουθήσει το σύστημα αυτό, μπορεί να το κλείσει όμως και το σύστημα ε, και υπάρχει πρόβλημα στην εναλλαγή πολλές φορές. Δεν είναι και κάτι εύκολο δηλαδή να εφαρμοστεί. Εμείς έχουμε διατυπώσει για την αυτοκινητοβιομηχανία και για τους δήμους και τις κοινότητες ένα αίτημα να υπάρξει δηλαδή εκπαίδευση για τους οδηγούς πάνω σε αυτή την τεχνολογία. Αλλιώς θα έχουμε καθυστέρηση στην εξέλιξη. Επίσης η πλήρη αυτοματοποιημένη οδήγηση είναι κάτι μακρινό σχετικά. Αν και υπάρχει τεχνολογία. Όμως θα πρέπει τα οχήματα αυτά να μοιραστούν τους δρόμους με τα συμβατικά οχήματα, όπως και με τους πεζούς και με άλλα ειδική χρήση ε, οχήματα. Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε 100% ασφάλεια και στην αυτόνομη οδήγηση, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν μεγαλύτερε απαιτήσει και δεν υπάρχει καμία ανοχή σε σφάλματα, ιδίω όταν μιλάμε για αυτοματοποιημένη οδήγηση. Πώς θα κυκλοφορήσουν τα οχήματα με αυτά τα διαφορετικά συστήματα ταυτόχρονα στους δρόμους. Εξού λοιπόν και θεωρούμε ότι τελικά είναι μια πρόκληση αυτό ε, για τη διαμόρφωση των ίδιων των ε, δήμων και των οδών. Θα πρέπει να υπάρξει διαχωρισμός της κυκλοφορίας ε, γιατί έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή η χάραξη των οδών είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο να ταυτόχρονα όλα αυτά τα οχήματα. Επίσης υπάρχει μια συζήτηση σε ό,τι αφορά τα δεδομένα και την πρόσβαση στα δεδομένα των ε, οχημάτων. Υπάρχει μια πίεση που έρχεται έξωθεν, έρχεται από κάποιους τρίτους, από πλατφόρμες και εμείς θεωρούμε, ξεκάθαρη απόψή μας, ε, ότι αυτός ναι μην είναι ένας νέος ε, τομέας, δραστηριότητας, αλλά προτεραιότητα έχει η ασφάλεια και μετά έρχονται τα δεδομένα. Εμείς θέλουμε να έχουμε ασφάλεια. Ε, δεν μπορεί να είναι τα, τα αυτοκίνητα σαν τα ε, τηλέφωνα, σαν τα smartphone, γιατί η ασφάλεια είναι πολύ σημαντικότερη σε αυτή την περίπτωση. Safety first λοιπόν στην περίπτωση της αυτοματοποιημένης πρώτης. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ ξεκάθαρη ήταν η δική σας τοποθέτηση. Θα παρακαλέσω τώρα τον κύριο Φαντεν Λίντεν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει και την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Good morning. Uh, on behalf of the Commission, I would... Καλημέρα. Στον όμορφο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση πριν δώσω το, το λόγο στον συνάδελφο. Η έκθεση φαίνεται να αναφέρει ότι τα Πλήρω αυτοματοποιημένα οχήματα θα είναι η εξέλιξη των συστημάτων CITS και δεν χρειάζεται πλέον η συνδεσιμότητα και συνεργασία. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί το CITS και τα συνδεδεμένα συστήματα θα συνεχίσουν να ισχύουν για όλα τα επίπεδα αυτοματοποίηση. Αντιθέτω, αν θέλουμε αυτά τα οχήματα να είναι 100% ασφαλή και πάντα, θα πρέπει να υπάρχει σύνδεση και συντονισμό των δράσεών του. Yes, good morning. Ευχαριστώ. Λαγκιόν ονομάζομαι τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξη. Συμπληρώνω αυτό που είπε ο συνάδελφο. Αρχικά, ε, θετική στήριξη προ την ανακοίνωση τη Επιτροπή του περασμένου Μαΐου. Ήθελα απλώ να πω ότι είναι μόνο η αρχή, το πρώτο βήμα των δραστηριοτήτων μα. Ήδη έχουμε περάσει στην υλοποίηση με την ε, με το σύστημα CITS προετοιμάζουμε ε, πρόταση κανονιστικού πλαισίου για αυτά τα οχήματα. Παράλληλα υπάρχει και το θέμα της πρόσβασης στα δεδομένα, τα οποία θίξατε αρκετή και εμείς συμφωνούμε ότι είναι πολύ σημαντικό και το επεξεργαζόμαστε. Θέλουμε λοιπόν να προετοιμάσουμε το έδαφος για πιθανές νομοθετικές ενέργειες. Όμως, όπως είπατε πολύ, πρέπει με μεγάλη προσοχή να εξετάσουμε τις επιμέρους επιλογές. Ήδη έχουμε αρχίσει όμως και θέλουμε να είναι έτοιμο αυτό το στάδιο στην, για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλος, είπατε ότι χρειαζόμαστε νομοθεσία. Έχω καλά νέα για εσά. Το επόμενο σημείο στην μέσα διάταξη είναι ακριβώς νομοθεσία κανόνες ασφαλείας για ε, τα οχήματα. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ανοίξουμε το δρόμο και για, τα αυτόνομα, για την αυτόνομη οδήγηση και σας καλούμε να σημειώσετε πρόοδο σε αυτό το φάκελο. Γιατί προβλέπει και ε, κανόνες ασφαλείας για αυτά τα οχήματα. Κάτι τελευταίο και σημαντικό, ο ανθρώπινος παράγοντας. Ναι, και εδώ έχουμε περάσει την υλοποίηση της ανακοίνωσης του τελευταίου περασμένου Μαΐου. Χθες η κυρία Μπούλς διοργάνωσε εκδήλωση για τον αντίκτυπο της αυτόνομης οδήγησης ε, στις θέσεις εργασίας. Απλώς θέλω να επισημάνω ότι έχουμε ήδη ξεκινήσει ε, τις εργασίες μας και σε αυτόν τον τομέα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι καλό που πριν από λίγο καιρό εγκρίναμε και το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Είναι η βάση για το μέλλον. Η ψηφοφορία... Α, ναι, όχι. Αύριο λοιπόν θα γίνει ψηφοφορία. Αλλά ίσως θα ήταν καλό να μας κάνει μία σύνοψη ο εισηγητής μας. Βίμ, πώς αντιδράς σε αυτά που άκουσες από τους συναδέλφους και από την Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Άκουσα και σημείωσα όλα τα σοφά λόγια των σκιωδών εισηγητών και υπολείπων συναδέλφων. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή για την έκθεσή της. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δύο γενικές διευθύνσεις, η DG Grow και η DG Tran, μας μίλησαν. Ελπίζουμε γρήγορα να φτάσουμε σε αυτή την νομοθεσία. Πρέπει να προσέξει η Ευρώπη να μην ε, μείνει πίσω, γιατί η Κίνα και οι Ηνωμένε Πολιτείε κινούνται πολύ γρήγορα. Πρέπει να περάσουμε στην πράξη και όχι απλά να μιλάμε. Ευχαριστώ. Ναι, είναι ένα πολύ αποφασιστικό θέμα ο ανταγωνισμός με Κίνα και είπα. Πριν προχωρήσουμε, αν με επιτρέπετε, θα ήθελα να καλωσορίσω την ε, δική μου ομάδα επισκεπτών από τη Θουριγγία. Είναι αρμόδιοι για logistics, ε, για τα ταξί, για τα πάντα. Ε, ό,τι έχει να κάνει με, την, με τον τομέα των μεταφορών και περνάμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης που έχει να κάνει με τι απαιτήσει έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων ρημουλκουμένων και συστημάτων κατασκευαστικών και χωριστών τεχνικών ομάδων όσον αφορά τη γενική ασφάλεια και την προστασία των επιβατών των οχημάτων και του ευάλωτου χρήστη τη οδού για την τροποποίηση του κανονισμού του 2018, Γενικού Κανονισμού για την Ασφάλεια. Η είναι η καθήλυνα αρμόδια ε, Τούν είναι η και εμείς ε, γνωμοδοτούμε για την ε, Επιτροπή ΙΜΚΟ. Ο Ματέις Φαν Μίλτεμπουργκ είναι ο συντάκτης της γνωμοδότησης και θα πρότεινα λοιπόν να του δώσουμε το λόγο για να μας παρουσιάσει την γνωμοδότησή του. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χθε είχαμε μια πολύ επικοδομητική συνάντηση των σκιωδών για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ του συναδέλφου για την ε, συνεργασία και ε, τη συμβολή του. Ε, η εξέβριση κοινού τόπου δεν είναι εύκολη, ιδίω ε, αν σκεφτείτε ότι έχουμε συνολικά 191 τροπολογίε, ε, κάποιε φορέ και αντίθετε μεταξύ του. Όμω είμαι πεπισμένο ότι θα έχουμε μια πολύ καλή γνωμοδότηση που θα δώσουμε στην ΙΜΚΟ. Έτσι κι η βελτίωση τη ασφάλεια στου Ευρωπαϊκού Δρόμου είναι ε, βασικό μέλημα τη επιτροπή μα. Θα ήθελα να επισημάνω ορισμένα από τα βασικά ζητήματα και δικαιβεύματα εδώ. Ε, θεωρώ ότι τα μέτρα ασφαλείας των οχημάτων που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν σημαντικές προεκτάσεις για την ασφάλεια στο δρόμο και δεν θα πρέπει να τα παίρνουμε ελαφρά. Όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτελεί σημαντική πρόοδο για την αυτόνομη οδήγηση, χαρακτηριστικά όπως ε, ε, τα συστήματα ε, που προειδοποιούν τον οδηγό όταν αλλάζει λωρίδα και διάφορα άλλα τέτοια συστήματα που υπάρχουν ήδη στην αγορά και νομίζω ότι πρέπει να τα υποστηρίζουμε να υποστηρίζουμε αυτές τις προδιαγραφές για λόγους ασφαλείας. Γι' αυτό και θα πρέπει να είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί σε σχέση με ορισμένες τροπολογίες που λένε ότι πρέπει να έχουμε και τη δυνατότητα εύκολα να απενεργοποιούμε αυτά τα χαρακτηριστικά. Ε, εκεί είμαι επιφυλακτικός γιατί πάλι τίθεται ζήτημα ασφαλείας. Θα δούμε όμως και στους συμβιβασμούς. Θεωρώ ότι ορισμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας όπως ε, ο καταγραφέας ε, συμβάντων ή ατυχημάτων θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά σε όλα τα οχήματα. Να μην εξαρτάται από το όχημα, τον τύπο ή τα, αν είναι πολυτελές ή όχι. Μετά θα πρέπει να ξεχνάμε και την προστασία δεδομένων, ιδίω ό,τι αφορά τον ε, καταγραφέα ατυχημάτων. Έχω εισαγάγει μια σειρά τροπολογίες για αυτό το ζήτημα και ελπίζω να βρούμε ευρεία συνένεση στους συμβιβασμού. Τέλος. Το Blind Spot Information System. Όπως ε, εισήχθη ε, σε κάποιες τροπολογίες. Αυτό το πρώτο λοιπόν αυτό το σύστημα είναι κάτι το οποίο αναλύει και αναφέρει αναλυτικά και διεξοδικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή της, στην πρόταση της μάλλον. Γι' αυτό θεωρώ ότι η εισαγωγή του Turning Assistance είναι περιττή. Όμως εδώ θα ήθελα ορισμένες διευκρινήσεις ή επιβεβαίωση της άποψής μου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να ξέρουμε αν ήδη περιλαμβάνεται στην πρόταση της Κομισιόν όπως εγώ νομίζω ή αν πρέπει όντω κάτι να προσθέσουμε για να το διευκρινίσουμε και φυσικά δεν θα έχω πρόβλημα σε αυτήν την περίπτωση ε, να βρούμε ένα συμβασμό. Ω Επιτροπή Τραν είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και φιλόδοξη αλλά και ρεαλιστική γνωμοδότηση για να δώσουμε στον κλάδο τον απαραίτητο χρόνο να καινοτομήσει και να επενδύσει. Όμως, από την άλλη, δεν πρέπει να ξεχνάμε τη δυνατότητα εισαγωγή αυτών των χαρακτηριστικών ασφαλείας για να βελτιώσουμε τελικά την ασφάλεια στους ε, δρόμους στην Ευρώπη. Είμαι ε, αρκετά αισιόδοξο ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Έχουμε και λίγο παραπάνω χρόνο γιατί η ψηφοφορία στην ΕΜΚΟ θα γίνει στις αρχές της επόμενης χρονιάς. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να αναβάλουμε την ψηφοφορία στην Επιτροπή μας εδώ μέχρι τις 10 Ιανουαρίου. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχω πει και στους σκιώδεις εισηγητές για να επεξεργαστούμε περισσότερο τις συμβαστικές τροπολογίες. Παρότι δεν είναι πάντα εύκολο, γιατί υπάρχουν τρει τροπολογίε μόνο και μόνο για τη διαγραφή ενό χαρακτηριστικού ασφαλεία που εγώ θεωρώ σημαντικό. Εκεί λοιπόν είναι αδύνατον να βρούμε συμβασμό και θα περάσουμε στην ψηφοφορία για να δούμε τι θα γίνει. Όμω συνολικά ε, είμαι ικανοποιημένο από την εξέλιξη των πραγμάτων και θα αξιοποιήσουμε και τον επιπρόσθετο αυτόν χρόνο ε, για να πετύχουμε ακόμα μερικέ ε, παραπάνω συμβαστικέ προτάσει. Ευχαριστώ πολύ. Προσβλέπω στη συνέχιση τη συνεργασία με του κοιότητε αυτή την ε, Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Φαμίλτεμπορκ. Περνάμε στους σκιώδεις εισηγητές. Εκ μέρους του ΕΛΚ είμαι εγώ, ο σκιώδης εισηγητής. Ξεκινώ λοιπόν εγώ. Θέλω να ευχαριστήσω ε, για τις συμβιβαστικές προτάσεις, ε, για την γνωμοδότηση ε, των συντάκτη μας και ζητώ συγγνώμη, αλλά θα πρέπει να φύγω για τις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 Βρυξέλ, μάλλον από τις Βρυξέλλες και δεν θα είμαι εδώ. Πάντως είμαστε πολύ καλά ε, εκπροσωπημένοι και θέλω να ευχαριστήσω που έλαβε ο κύριος Φαμίλτεμπορ και υπόψη τις δικές μας προτάσεις. Όπως είπατε, λάβατε 191 τροπολογίες ε, και έχετε κάνει κάποιες συμβαστικές προτάσεις. Ε, όπως βλέπω εγώ, καλύπτονται όμως μόνο 27 ουσιαστικά από τα θέματα και υπάρχουν και κάποιες ταυτόσιμες τροπολογίες. Είχαμε ε, συνάντηση ε, σχεδόν και στην επόμενη που θα κάνουμε θα προτείνω να συμπεριληφθούν και άλλες από τις ε, τροπολίες που έχουν ήδη συμπεριληφθεί στις συμβιβαστικέ και θα ζητήσω να υπάρξουν και νέες συμβιβαστικέ προτάσεις. Ε, υπάρχουν κάποια επίμαχα θέματα. Νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε από αυτόν ε, μια κοινή τοποθέτηση. Τουλάχιστον αυτό θα προσπαθήσουμε και όχι να εστιάζουμε από την αρχή στην πρόταση της Κομισιόν και να μένουμε εκεί. Αν και η πρόταση αυτή είναι καλή φετηρία. Θεωρώ ότι είναι καλή αυτή η πρόταση της Κομισιόν γιατί ουσιαστικά περιλαμβάνει αυτά τα οποία είχα συμπεριλάβει και εγώ στη δική μου έκθεση πρωτοβουλίας πριν από 1,5 χρόνο. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν θέματα ε, που καλό είναι να βελτιωθούν ε, περαιτέρω στην πρόταση της Κομισιόν και υπάρχουν και κάποια επίμαχα από τον οποίο καλό είναι να βρούμε μια κοινή λύση. Έχω λοιπόν καταθέσει τις προτάσεις μου στο πλαίσιο της ε, και ε, πρόταση των συγητών και η συνεργάτη μου θα παρουσιάσει ε, στην επόμενη συνεδρίαση των σκιωδών που δεν μπορώ εγώ να παραστώ τις ε, νέε μου αυτές προτάσει. Θα πρέπει λοιπόν από κοινού να δούμε πώς θα προχωρήσουμε, αν μπορούμε να καταθέσουμε μια κοινή πρόταση σε ό,τι αφορά την πραγματική βελτίωση της οδικής ασφάλειας διότι νομίζω ότι αυτό είναι ο κοινό μα στόχο και κατά την άποψή μου θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να τον πετύχουμε, γιατί είναι σημαντικό για του πολίτε αυτό και το ξέρετε. Βέβαια, όποιο ε, αγωνίζεται μπορεί να κερδίσει, ε, μπορεί και να χάσει, αλλά όποιο δεν αγωνιστεί είναι χαμένο από χέρι. Και εμεί αυτό θέλουμε να κάνουμε, να αγωνιστούμε για την οδική ασφάλεια, για του πολίτε μα, άνδρε και γυναίκε. Ευχαριστώ. Και τώρα εκ μέρους ε, Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ε, η Όλγα Σενιάλοβα είναι εδώ η συγγήτρια Ισκιώδης. Παρακαλώ Όλγα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι είχαμε την συνάντηση των σκιωδών. Εξετάσαμε όλες τις ε, πιθανές συμβιβαστικές προτάσεις και διαλευκάναμε και κάποια θέματα Είχαμε λάβει πολλές τροπολογίες και έπρεπε να διευκρινιστούν κάποια πράγματα από αυτόν. Είναι τροπολογίες που πολλές φορές διαφέρουν πολύ μεταξύ τους. Δεν ήταν και εύκολο λοιπόν να καταλήξουμε σε κάποιες συμβαστικέ προτάσεις. Και σίγουρα έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας. Πάντως ε, έχουμε συμφωνήσει σε κάποιες προσεγγίσεις. Παραδείγματος χάρη το θάλαμο, τι μορφή θα πρέπει να έχει. Ε, και σίγουρα στόχος είναι να βελτιωθεί ορατότητα των οδηγών για να έχουν καλύτερη ιδέα για το τι γίνεται γύρω από το όχημά τους. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, είναι μια καλή συμβαστική πρόταση. Στηρίζω επίσης μια άλλη συμβαστική πρόταση για το είδος των ελαστικών. Σε ό,τι αφορά τις δοκιμές που γίνονται ε, ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης ή η καταγραφή δεδομένων συμβάντων ή ατυχήματος ή ατυχημάτων. Θα πρέπει αυτό το θέμα τη καταγραφή των δεδομένων, είναι πολύ σημαντικό, να διευκρινιστεί όχι μόνο σε την προστάση των δεδομένων, αλλά και την αποτελεσματικότητα αυτού του μηχανισμού. Συμφωνήσαμε επίσης να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας ε, πάνω στις συμβιβαστικές προτάσεις ε, και να συμπεριλάβουμε και άλλες τροπολογίες αυτές τις ήδη σε Πολύ καλή συνεργασία και με τον Πρόεδρο και νομίζω ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια θέση που πραγματικά θα μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία και να περιληφθεί η δική μας νομοδότηση στην, αρμόδια, στην έκθεση αρμόδιας επιτροπής της Επιτροπής ΣΥΜΚΟ δηλαδή. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ την Όλα Σενιάλοβα. Από το ECR, από του ε, συντηρητικού ε, δεν βλέπω τον κύριο ε, εσείς κύριε Λούντγκρεν, πως θα θέλετε κάτι να πείτε. Ναι, βεβαίω, κάτι μπορώ να πω. Δεν είμαι οπαδός του ηλεκτρονικού εξοπλισμού που θα αφαιρέσει την ευθύνη του οδηγού Κατά τη γνώμη μου θα ήταν πολύ καλύτερο να εκπαιδεύονται οι οδηγοί ώστε να είναι καλύτεροι οι οδηγοί γιατί όση τεχνολογία και αν βάλουμε στα αυτοκίνητα, στον κόσμο του οδηγού δεν θα βοηθήσει γιατί και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός δυσλειτουργεί από καιρό εις καιρόν. Κοιτάξτε έναν κομπιούτερ. Αν ένας κομπιούτερ ήταν αυτοκίνητο θα είχαμε ε, ατυχήματα όλη την ώρα γιατί ξαφνικά σταματάει και πρέπει να το σβήσουμε και να το ξανα ε, ανάψουμε και θα εξαρτώμεθα δηλαδή από τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό στο αυτοκίνητο να αναλάβει να λύσει το θέμα, το πρόβλημα. <clears throat> Όπως γνωρίζετε είμαι και οδηγός φόρμουλας. Ο οδηγός είναι αυτός που, που σώζει την κατάσταση όταν ε, προκύψει πρόβλημα σε κάποιο αγώνα ράλι. Τελικά λοιπόν πρέπει να εκπαιδευτεί ο οδηγό ώστε να είναι καλύτερο οδηγό. Γιατί ειλικρινά υπάρχουν αρκετοί γρήγοροι οδηγοί. Το βλέπω καθημερινά. Και όση τεχνολογία και να βάλει στα αυτοκίνητά τους δεν θα βοηθήσει γιατί απλώς δεν ξέρουν να οδηγούν σωστά. Όπως σας είπα είναι ένας, όπως ένας υπολογιστής. Εάν κανείς δεν τον χειρίζεται με το σωστό τρόπο, καλύτερα να χρησιμοποιεί μολύβι και χαρτί. Το ίδιο λοιπόν ισχύει και για τους οδηγούς. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Λούντγκρεν. Όλοι ξέρουν, όλοι νομίζουν ότι είναι οι καλύτεροι οδηγίες. Λέτε δεν είστε. Τέλος πάντων δεν είναι σύνηθες κύριος Κράμερ, Μιχαλ Κράμερ τώρα, σκιώδης του Πρασίνου. Πρασίνους. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή αλλά και τους σκιώδης εισηγητές. Ήταν μια πραγματικά πολύ καλή συζήτηση και ο σκιώδης εισηγητής ε, του ε, ΕΛΚΑ εκπροσωπήθηκε από την συνεργάτη δάτου στην προηγούμενη συνάντηση. Πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία εμεί ω πράσινοι θέλουμε να αναφέρουμε. Πρώτα απ' όλα σε ό,τι αφορά την υποβοηθούμενη οδήγηση, ότι είναι ένα σύστημα που μπορεί να εφαρμόζεται μόνο στα νέα οχήματα. Εμεί θέλουμε να υπάρχει πανεξοπλισμό ε, των παλαιότερων οχημάτων, γιατί αυτό μπορεί να ε, πάρει χρόνια και πρέπει να προστατεύσουμε τον κόσμο από βαρύ τραυματισμού και άλλα ατυχήματα. Καλό λοιπόν να μπορεί να τοποθετηθεί εκ των υστέρων ε, ο εξοπλισμός αυτός. Τώρα τα όρια ταχύτητας ε, σε όλα τα ε, οχήματα και αυτό είναι σωστό. Αν υπάρχει υπέρβαση του όριο ταχύτητας θα πρέπει να δίνεται ένα σήμα, να ενημερώνεται ο οδηγός. Το θέμα είναι κλείνει αυτός ο μηχανισμός. Εμείς θα θέλαμε το όριο ταχύτητας να μπορεί κάποιος οδηγός να το υπερβεί. Μπορεί να υπάρχουν ε, περιπτώσεις ε, που εγώ θα επιταχύνω ταχύτητα για να γλιτώσω ένα ατύχημα, μια σύγκρουση για παράδειγμα, οπότε μπορώ να τον κλείσω ίσως το μηχανισμό. Το θέμα είναι τι γίνεται αν είναι μόνιμα κλειστό αυτό το σύστημα. Μήπως τελικά αυξηθεί ο αριθμός των τραυματιών και των ε, νεκρών. Γι' αυτό εγώ λέω θα πρέπει να είναι πολύ ε, σαφές το όριο, να μην μπορεί κανείς να υπερβεί ένα συγκεκριμένο όριο και τώρα αν ε, ξέρει ότι ε, αυτό δημιουργεί πολύ περισσότερους ε, κινδύνους ε, μπορεί ίσως να το κλείνει για λίγο για να περάσει ένα φορτηγό κτλ. Αλλά καλό είναι να μην ε, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ό,τι αφορά τον έλεγχο κατανάλωσης αλκοόλ, προς το παρόν προβλέπεται για τα βαρέα οχήματα. Εμείς όμως το θέλουμε για όλα. Γιατί ο κίνδυνος από την κατανάλωση αλκοόλ στο τιμόνι είναι πολύ μεγάλος. Είναι η πιο συχνή πρόκληση ε, ατυχήματος. Ε, και ακόμα και ο οδηγός ταξί είναι επαγγελματίας δεν ε, πρέπει μόνο τους φορτηγατζίδες αλλά και τους αξιτζίδες ε, να τους ελέγχουμε. Επίσης το λεγόμενο Doring είναι μια νέα τεχνολογία την οποία θέλω να αναφέρω που σημαίνει οι περισσότεροι ποδηλάτες ε, κινδυνεύουν όταν ανοίγει την πόρτα ο οδηγός του αυτοκινήτου την ώρα περνάνε. και Κάποιοι μπορεί να είναι στο κινητό τους ε, μπροστά και να μην προσέχουν ή να μην βλέπουν τέλος πάντων ποιος έχει από πίσω. Το ντόρινγκ λοιπόν το άνοιγμα της πόρτας που χτυπάει έναν ε, ποδηλάτη είναι ένας μεγάλος κίνδυνος ε. Ε, δεν ξέρω αν γίνεται να υπάρχει ένα σύστημα που να μην ανοίγει πόρτα. Νομίζω στην ε, Ολλανδία ε, δεν μπορεί κανείς να αλλάξει παραδείγματο χάρη χέρι για να ανοίξει. Πρέπει πρώτα να ελέγξει κτλ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες. Κάποιοι κατασκευαστές έχουν, αλλά μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ε, εξοπλίσει κάποια οχήματα με ένα τέτοιο σύστημα. Εγώ νομίζω όμως ότι θα αυξηθεί τεράστια η ασφάλεια. Το 40% των ατυχημάτων με ποδηλάτης είναι λόγω ανοίγματο πόρτας αυτοκινήτου. Έχουμε καταθέσει σχετική τροπολογία. Θα δούμε. Ε, θα συνεργαστούμε και με την Επιτροπή ΙΜΚΟ Καλό θα ήταν όμως νομίζω να υπάρξει μεγάλη πλειοψηφία που να υποστηρίζει την πρόταση αυτή. Πρόεδρο. ευχαριστώ τον κύριο Κράμερ. Νομίζω ολοκληρώσαμε το γύρο των σχεδόν εισηγητών. κυρία Γιάλα Σέντερ, ΝΕΣ, νομίζω ότι ήθελε το λόγο εσύ, ε, είσαι η μόνη από τους υπόλοιπους συναδέλφους, ε, παρακαλώ. πείτε το έχει ζητήσει το λόγο. Ναι, ναι, με συγχωρείτε, Πρόεδρε. Απλά ήμουν απασχολημένη και μελετούσα τον κατάλογο ψηφοφορία ε, για το Connecting Europe. Ακριβώ επειδή μας απασχολεί ακόμη αυτό το θέμα του Connecting Europe, δεν μπόρεσα να μελετήσω όλες τις προτάσεις και όλες τις τροπολογίες. Ε, οπότε μια ερώτηση έχω προς τον κύριο Φαν Μίλτεμπουργκ. Πρώτον, από ό,τι βλέπω, όλα όσα έχουν να κάνουν την προστασία δεδομένων, μηχανισμούς και επιπτώσεις, προβλέπονται μέσω ενός εγχειριδίου που θα γίνουν ε, πάρα πολύ τεράστια ε, ογκώδη τελικά αυτά τα εγχειρίδια. Οπότε εγώ λέω μήπως θα ήταν δυνατόν, αλλά δεν έχω δει και τις τροπολογίες όλες τουλάχιστον σε σχέση με το θέμα αυτό. Μήπως θα ήταν δυνατόν να υπάρχει ένα συμβόλαιο που να υπογράφουν. Κάποιες τέτοιες το κάνουν. Μία Αμερικανική συγκεκριμένα όχι ευρωπαϊκή, που όσους αγοράζουν τους βάζει να υπογράψουν ένα συμβόλαιο με όλα τα δεδομένα. Αυτό βέβαια δεν είχα κάνει τόσο με την προστασία, αλλά με τη χρήση των δεδομένων. Αλλά αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό για τους οδηγούς, έστω ε, μεταβατικά, να γνωρίζουν τι αγοράζουν, περί αυτού που πρόκειται ουσιαστικά να είναι ένα είδος ε, ε, πομπού ή δέκτη δεδομένων το αυτοκίνητο. Και επειδή ο κύριος Φαμίλτεμπουργκ είναι αντίθετος ε, με τροπολογία 10 λέει ε, τις δημόσιες αρχές, τις δημόσιες διοικήσεις να μπορούν να χρησιμοποιήσουν ανώνυμοποιημένα δεδομένα για το πώς να το πω Α, ναι, για τις στατιστικές, για τροχέα. Εγώ νομίζω ότι Ακριβώς το αντίθετο. Θα έπρεπε να τα χρησιμοποιούνται, αλλά να χρησιμοποιούνται αυτά ανώνυμο, ανώνυμα δεδομένα για ακριβώς τους σκοπούς αυτούς της δημόσιας ασφάλειας, πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος που να θέλει το λόγο. Πάμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γάμα Δέλτα ΓΡΟ. Πίτερ Πρόιτς. Έχετε το λόγο. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή κύριο Βαν Μούντενμπουργκ. για όλη την προσοχή που έχει δώσει στην πρωτοβουλία μας για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας μέσω της βελτίωσης της ασφάλειας οχημάτων. Κύριε Κόχ, πολύ ορθά αναγνωρίσατε ότι είστε μεγάλη πηγή έμπνευση για αυτή την πρόταση με την, με την έκθεση της πρωτοβουλίας. Με τα χαράς βλέπουμε ότι οι συζητήσεις ε, προχωρούν στο Κοινοβούλιο. Θα θέλαμε να σχολιάσουμε ορισμένα μόνο πράγματα. Πιο συγκεκριμένα, οι τροπολογίε που αφορούν συγκεκριμένες τεχνολογίες ή μάλλον μέτρα που προτείνουμε, για παράδειγμα το Intelligence Speed and Assistance σε ό,τι αφορά την υποβοηθούμενη ταχύτητα, μπορεί να σημαίνει ότι εναλλακτικά συστήματα, όπως ένας δείκτης που σας δείχνει το, την ταχύτητα, αντί του συστήματος που προτείνουμε εμείς, που κάπως συνεργάζεται με τον οδηγό, ότι θα έχει την ίδια αποτελεσματικότητα, αλλά αυτό δεν ισχύει. Το σύστημα που προτείνουμε εμείς έχει αντίκτυπο 17 έως 19% μείωσης του κινδύνου. Όταν αποδυναμωθεί το σύστημα μόνο σε ένα σύστημα πληροφοριών ε, ορίου ταχύτητας, ε, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Το Intelligence Speed Assistance που λέμε εμείς είναι το καλύτερο μέτρο που έχουμε. Ουσιαστικά περιορίζει μερικά χιλιόμετρα την ώρα, αλλά έχει τεράστιο αντίκτυπο σε ό,τι αφορά τον περιορισμό του κινδύνου και των ε, θανατηφόρων ατυχημάτων. Γιατί το όφελος αυτό ε, φτάνει κλιμακωτά σε όλα τα στάδια. Επομένω, να το διατηρήσετε αυτό, παρακαλούμε. Ακόμα εξετάζουμε τα ε, τα στοιχεία, τα δεδομένα, αλλά μιλάμε για εκατοντάδες, να μην σας πω χιλιάδες ζωές που θα σωθούν αν αλλάξουμε από το ένα σύστημα στο άλλο. Κατανοώ ότι υπάρχουν επιφυλάξει για την αξιοπιστία, τη διαθεσιμότητα του συστήματος. Τα συστήματα όμω υπάρχουν στην αγορά. Κάποιοι κατασκευαστές σημειώνουν μεγάλη ε, επιτυχία Στι δοκιμέ γύρω αν κάποιο παράδειγμα παίρνουν πολύ μεγάλη βαθμολογία. Κάποιε μελέτε, βέβαια ξέρω ότι λένε ότι υπάρχει ένα ποσοστό σφάλματος 10% σήμερα ή μάλλον πριν από μερικά χρόνια μάλλον. Αν εγώ στην έκθεσή μου ε, έπαιρνα 9 στα 10, μια χαρά χαρούμενος θα ήμουν. Είναι πολύ καλός βαθμός τα 9 στα 10. Και θα βελτιωθεί κι άλλο γιατί τώρα είμαστε στο 2018 ρεαλιστικά αν το δείτε. Αν δούμε το 2020-2022, θα υπάρχει υποχρεωτικά αυτό το χαρακτηριστικό στα νέα μοντέλα και μετά αργότερα θα είναι για όλα τα οχήματα. Ήδη έχει βελτιωθεί πολύ λοιπόν ε, η τεχνολογία. Και αυτά τα συστήματα έχουν να κάνουν και με τις πληροφορίες υποδομών. Μίλησαμε προηγουμένως για την αυτόνομη οδήγηση. Πιστέψτε με, και το αυτόνομο όχημα θα πρέπει να ξέρει την ταχύτητα. Είναι απολύτω απαραίτητο. Τα κάτι μελη λοιπόν δεν έχουν άλλη επιλογή από το να βελτιώσουν αυτέ τι πληροφορίε. Και το bonus εδώ είναι ότι το ΆΙΖΑ, το σύστημα το οποίο θα καταστήσετε υποχρεωτικό, θα λειτουργήσει πολύ καλύτερα από ό,τι σήμερα. Επομένως, σας παρακαλούμε να το λάβετε σοβαρά υπόψη. υπήρξαν και κάποιες άλλες παρατηρήσεις για τους κακούς οδηγούς. Ναι, ισχύει. Και το πακέτο που προτείνουμε εμεί σα προστατεύει και από αυτούς τους κακούς οδηγούς. Αν είναι, ας πούμε, κάποιος καλός οδηγός και διασταυρωθεί με έναν κακό οδηγό, αυτά τα συστήματα έχουν τη δυνατότητα να σας σώσουν τη ζωή. Το assistance system που σας πρότεινα προηγουμένως δεν είναι ένας μηχανισμός ε, Big Brother που θα σας παρακολουθεί και δεν θα σας επιτρέπει να πάτε παραπάνω με μεγαλύτερη ταχύτητα, αλλά θα σώσει πολύ περισσότερες ζωές. Θα ξέραμε μάλλον ότι αν σας προτείναμε αυτό θα έσωσε ακόμα περισσότερες ζωές, αλλά θα ήταν υπερβολικό. Γι' αυτό και εμείς δεν το προτείνουμε αυτό ε, κάτι δηλαδή το οποίο αυτομάτως θα σας ε, κόβει την ταχύτητα, είναι κάτι το οποίο συνεργάζεται με τον οδηγό και έτσι δεν ενοχλείται ο οδηγός. Και αν για κάποιο λόγο δεν υπάρχει το όριο ταχύτητας διαθέσιμο, έχουμε την ε, κλασική συμβατική οδήγηση. Όπως κάνετε τώρα, που βλέπετε ε, ποιο είναι το όριο ταχύτητας και το τηρείτε. αυτός είναι ο μηχανισμό υποβοήθησης λοιπόν στην ταχύτητα. Εμείς όμως δεν θέλουμε να έχουμε υποχρεωτικές ε, τέτοιες λειτουργίες υποβοήθηση της οδήγησης. Δεν θα είναι adaptive cruise control. Είναι ένα σύστημα ε, καταπήγοντος φρένου της τελευταίας στιγμής. Βέβαια θα τα δούμε και στην πορεία γιατί χρησιμοποιούν τους ίδιους αισθητήρε και για την ε, παραμονή στην ίδια λωρίδα. Μιλάμε και για τον αντίστοιχο μηχανισμό emergency ε, lane keeping ε, assistance. Αν δείτε με προσοχή την ε, πρόταση, πρόκειται μόνο για τις περιπτώσεις όπου επίκειται ατύχημα. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε υποχρεωτικά κάποια στοιχεία ε, ευκολίας, αν θέλετε, που θα οδηγεί τους οδηγούς στον εφησυχασμό. Και τέλος, το dooring, αυτό που ανοίγουν τις πόρτες και χτυπάνε τους ποδηλάτες. Το έχουμε εξετάσει, δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε τα στοιχεία, κατά πόσο δηλαδή είναι 40% το ποσοστό των ατυχημάτων που προκύπτουν ε, με τα ποδήλατα είναι μια νέα τεχνολογία. Ξέρουμε ότι κάποιοι κατασκευαστές προσπάθησαν να λαντσάρουν κάτι στην αγορά, αλλά δεν ήταν αξιόπιστο, ούτε αρκετά γρήγορο, ήταν και πολύ περίπλοκο. Γι' αυτό θεωρήσαμε ότι απαιτείται και άλλη δουλειά πριν ε, κάνουμε μια τέτοια πρόταση. Δεν το στηρίζουμε ακόμα. Και τέλος, ζήτησε ο κ. Βαρμίλτον να επιβεβαιώσουμε ότι το Turning Assistant ή το Blind Spot Information System υπάρχουν στην πρόταση. Πράγματι, η αρχική πρόταση εξετάζεται δύο πράγματα ξεχωριστά. Πρώτον, το turning assistance, το blind spot information, δηλαδή όταν το φορτηγό ε, στρίβει και χτυπάει ένα ποδηλάτι κατά κύριο λόγο. Και στο ίδιο άρθρο έχουμε τα ατυχήματα όπου ξεκινάει σιγά σιγά το ε, αυτοκίνητο όταν οι πεζοί, συνήθω παιδιά, ε, διασχίζουν τον δρόμο, είναι πολύ κοντά μας το ε, όχημα, γι' αυτό δεν τα βλέπει ο οδηγό. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα δύο στοιχεία σε αυτά τα άρθρα. Επιβεβαιώνουμε λοιπόν ότι καλύπτονται αυτά τα δύο στοιχεία σε αυτά τα άρθρα. Θέλουμε λοιπόν αυτή η τροπολογία να υιοθετηθεί, όπως προτείνει ο εισηγητής. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Εσείς κύριε Κράμερ, αν μπορώ, πριν ξαναπάρει το λόγο εισηγητής, μια σύντομη ερώτηση για τον Ντόρινγκ, για να σας δώσω πληροφορίες. Η Bild έχει ένα άρθρο για τη Mercedes. Ότι σας φροντίζει. Ότι φροντίζει τους ε, ποδηλάτες. Και υπάρχουν και άλλα άρθρα. Η τεχνολογία σώζει ζωές. Και για να γίνει αρθρό σημαίνει ότι έχει προηγηθεί κάποια εξέλιξη. Άρα και η Mercedes βάζει τέτοια συστήματα και άλλε. Δεν καταλαβαίνω γιατί λέει τότε η Κομισιόν ότι πάμε πολύ γρήγορα και δεν μπορούμε να πάμε τόσο γρήγορα. Αφού υπάρχουν άρθρα που το λένε. Καλό θα ήταν να το εφαρμόσουμε αυτό το σύστημα γιατί θα σώσει πραγματικά ζωέ. Πρώτα, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την προσθήκη κύριε Κράμερ. αυτό που είπατε για ε, την ε, ευφύ υποβοήθηση ε, σε ό,τι αφορά την ταχύτητα, την ενημέρωση για το ότι κτλ. κτλ. Τα σημείωσα και δίνω το λόγο στον κύριο Φαν Μίλτεμποργκ για να κλείσει. Yeah, thank you, Chair. Very shortly. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, με συντομία. Φυσικά, εκεί που μπορούμε να βρούμε κοινό τόπο για περαιτέρω συμβαστικέ τροπολογίε, θα το πράξουμε. Και χθε, για παράδειγμα, εξετάσαμε και, την... και διάφορε advanced restriction recognition. Κάποιοι συνάδελφοι ήθελαν να το διαγράψουν για πολλού λόγου. Κάποιοι συνάδελφοι έχουν επιφυλάξει σε ό,τι αφορά την προστασία δεδομένων και ιδιωτικότητα. Οπότε συμφωνώ με αυτό το σημείο και θα εξετάσω ε, αυτή την πρόταση, ίσως καταθέσω άλλη συμβαστική τροπολογία για την προστασία δεδομένων, όπως είπε η κυρία Γιάλα Σέντερ. Ίσως θα ήταν καλύτερα να σας στείλω το νέο κείμενο των συμβαστικών τροπολογιών. Εκεί, α πούμε, λέμε ότι οι κατασκευαστές θα διασφαλίσουν ότι δεν θα είναι ιχνηλάσιμοι αυτή ε, αυτοί οι μηχανισμοί ε, καταγραφής ατυχημάτων Νομίζω ότι όλα αυτά συνδέονται και με τη συζήτηση για το e-call. Θα καταλήξουμε σε κάποιο συμβασμό για το event data recorder. Αν κατάλαβα καλά, θέλετε να χρησιμοποιηθούν δεδομένα και για μεμονωμένες έρευνες μετά από ένα ατύχημα. Εδώ είμαστε λίγο πιο επιφυλακτικοί. Να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα για ερευνητικούς σκοπούς, αλλά ευρύτερα, όχι για επιμέρους έρευνες μετά από ένα τύχημα. Όπως και να έχει, θα αξιοποιήσουμε τον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας για να βρούμε επιπρόσθετες συμβαστικές τροπολογίες για να ψηφίσουμε στις 10 Ιανουαρίου. Αλλά πρέπει να έχουμε και κατά νου ότι κάποιες φορές Έχουμε πολύ διαφορετικές ε, τροπολογίες και παρότι πάντα είμαι διατεθειμένος ε, να τα συζητήσω για να βρω επιπλέον ε, συμβαστικές τροπολογίες, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να στείλουμε και κάτι, μια γνωμοδότηση στην Ήμικο που να έχει και κάποιο νόημα. Να πούμε λοιπόν ξεκάθαρα τι θέλουμε, αν θέλουμε αυτά τα συστήματα ή όχι. Πρέπει αυτό να είναι σαφές. για λόγους ε, ποιότητα της νομοδότησης που θα στείλουμε στην ΕΜΚΟ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φανλούκεμπουργκ. Το 92% των τροχαίων οφείλονται σε ανθρώπινο λάθο. Άρα σίγουρα χρειάζεται καλύτερη οδήγηση. Και καλό είναι βέβαια να υπάρχουν και τα συστήματα που έστω και το τελευταίο δευτερόλεπτο μπορούν να βοηθήσουν ε, τους οδηγούς να αποφύγουν επικίνδυνες καταστάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ψηφίσουμε α, στις 10 Ιανουαρίου την έκθεσή σου αυτή και προσβλέπω και στη συνέχεια της καλής μας συνεργασίας και τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόθεση της δικαιοσύνης και της διαφάνειας. Κλάουντια Ταπαρδέλ. Σας ευχαριστώ. Είμαι πολύ ικανοποιημένη γιατί μπορώ να σας πω γιατί μετά από τις συζητήσεις με τους σκιώδεις ηγετές καταφέραμε ε, ε, ισορροπημένες ε, συμβιβαστικές τροπολογίες. Η έκθεση αυτή λοιπόν θα είναι ισορροπημένη γιατί συγκέντρωσε την συνεργασία όλων των σκιωδών εισηγητών και οι οποίοι έδειξαν ιδιαίτερα θετικό πνεύμα ώστε να φτάσουμε σε συμβιβαστικές λύσεις. Ε, η έκθεση λοιπόν είναι ισορροπημένη, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει τη διαφάνεια για τους παρομηθευτές υπηρεσιών, τους καταναλωτές και τους καταναλωτές επιγραμμικά. Ελπίζω λοιπόν πως θα μπορέσουμε να εγκρίνουμε όλες αυτές τις συμβιβαστικέ. Ε, η νέα είναι πρόοδος. Γιατί? Γιατί ορίσαμε σημεία κλειδιά, δηλαδή τη διαφάνεια. Τι σημαίνει αυτό? ότι οι πλατφόρμες οφείλουν να ενημερώνουν τον ε, προμηθευτή για το κατά πόσο χρησιμοποιούν ε, συγκεκριμένες διόδους για να ε, προσφέρουν υπηρεσίες και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά, ε, αυτά τα κανάλια επικοινωνίες. Θεωρήσαμε πως είναι καλό να χρησιμοποιηθουν αυτα τα καναλια επικοινωνιας θεωρησαμε πως ειναι καλο να υπαρχει μια περίοδος 15 με 30 ημερών πριν να μπορέσουν να κάνουν οποιαδήποτε αλλαγή. Η περίοδος κοινοποίησης δεν μπορεί να ισχύσει όταν η αλλαγή γίνεται άμεσα, γιατί έτσι ο νόμος μπορεί να παραβιαστεί από το προμηθευτή. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν ε, πρέπει οι ε, εκθέσεις να δίνονται αμέσως. Οι εμπόροι μπορεί να διαπραγματευτούν το φόρο που έχουν πληρώσει για αυτές τις, σε αυτές τις πλατφόρμες και εκεί έχουν ένα δικαίωμα διαπραγμάτευσης και έτσι εγγυόμαστε μια ισορροπία ανάμεσα στις, στα διάφορα εμπλεκόμενα μέρη. Όσον αφορά τη συμβιβαστική 12, είναι εξίσου σημαντική γιατί καλύπτει το σύστημα ταξινόμησης των προμηθευτών στις πλατφόρμες παροχής υπηρεσιών. Οι παράμετροι αυτές θα πρέπει να ε, εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις για τους παρόχους των υπηρεσιών και οποιαδήποτε περαιτέρω αλλαγή θα πρέπει να κοινοποιείται έγκαιρα στους προμηθευτές, δεδομένου ότι αυτό τα όλα είναι πάρα πολύ σημαντικά για τους παρόχους των υπηρεσιών αλλά και για τους καταναλωτές γιατί αυτοί είναι που λαμβάνουν τις σημαντικές αποφάσεις ε, ε ταξινόμησης. <coughs> και καταχώρησης. Για τα πρώτα αποτελέσματα που βγαίνουν όταν κανείς κάνει μια αναζήτηση online, θα πρέπει η κατάταξη αυτή να γίνεται με διαφανή τρόπο και χωρίς να γίνονται διακρίσεις. Κάτι ακόμα το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό και για το τουρισμό, ε, και ως προς αυτό είμαι ευτυχής που μπόρεσα να έχω τη βοήθεια διαφόρων πολιτικών ομάδων δεδομένων των αποκλήσεων των απόψεων για αυτά τα θέματα. Οι ε, πλατφόρμες ε, θα πρέπει να προσφέρουν στον καταναλωτή άλλες υπηρεσίες και εδώ θέλω να παραθέσω το ρήτρα του πιο ευνοούμενου κράτους. Εγώ θα ήθελα να υπάρχει να ελεύθερη αγορά και ελεύθερος ε, θεμητός ανταγωνισμός. Ε, άρα λοιπόν ξεκινάμε από την αρχή ότι όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών θα μπορούν να προσφέρουν ε, υπηρεσίες με διά... από όλα τα διαφορετικά μέσα που υπάρχουν. Ας πούμε, ο τουρισμός αυτό θα πρέπει να ωφελήσει τον καταναλωτή και άρα ο καταναλωτής θα έχει τη δυνατότητα να έχει την καλύτερη προσφορά στην καλύτερη τιμή. Και για τη συμβιβαστική 8 εγγυόμαστε το γεγονός ότι οι επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να προσφέρουν μη διακριτική μεταχείριση όσον αφορά την εισαγωγή ορισμένων κυρώσεων απέναντι στους προμηθευτές. Ας πούμε, η ακύρωση συμβολέου, η αναστολή, η επιστροφή, η αποζημίωση κτλ. Οι πλατφόρμες δεν μπορούν από τη μια μέρα στην άλλη να διακόπτουν συμβάσεις διαγράφοντας την ύπαρξη ενός παρόχου ε, χωρίς να ε, το αιτιολογούν και χωρίς αυτός να έχει ενημερωθεί εκ των προτέρων. Είναι σημαντικό λοιπόν ότι εδώ έχουμε να κάνουμε πολύ ευαίσθητα θέματα για την ψηφιακή οικονομία και νομίζω πως τελικά είχαμε μια ισορροπημένη ε, προσέγγιση για όλους. Οι πλατφόρμες, ο ε, ε, καταναλωτής ε, νομίζω πως θα ωφεληθούν. Με ενδιαφέρον περιμένω τη γνώμη σας και ελπίζω πως θα βοηθήσετε με την θετική σας ψήφο για αυτή την έκθεση. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Ταπαρδέλ. Ισκιώδης τώρα. Από τις διάφορες πολιτικές ομάδες, ο Βίμ. Θα πάρεις εσύ το λόγο μέρος του ΕΛΚΑ. Σου δίνω το λόγο λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορούσε να είναι εδώ η, η να πάει να ψηφίσει σε μια επιτροπή. Οπότε αναλαμβάνω εγώ το ρόλο να ευχαριστήσω ε, τη σκιοδησηγήτρια η πλατφόρμες αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικές. Πάνω από ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις ε, στην Ευρώπη χρησιμοποιούν. Και ε, πρέπει να δημιουργηθεί ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ιδίως για τις μεταφορές. By online και επηρεάζουν οι επιγραμμικές πλατφόρμες και η ψηφιακή οικονομία. Υπάρχουν πολλές ΜΜΕ που θα μπορούσαν να ωφεληθούν από σαφέστερους πιο διαφανείς κανόνες και αυτό το επίπεδο του ανταγωνισμού δεν είναι εύκολο να ρυθμιστούν όλες αυτές οι επιγραμμικές πλατφόρμες γιατί εμπλέκονται πάρα πολύ διαφορετικοί τομείς όμως αυτός, ο στόχος μας είναι να βρούμε ισορροπία. Η πρόταση της Κομισιόν είναι καλή, αλλά οι συμβιβαστικές τροπολογίες θα καταστήσουν ακόμα μεγαλύτερη την ισορροπία αυτής της προσέγγισης. Η συγκίτρια κυρία Κλάουντια Ταπαρδέλ έχει κάνει πολύ καλή δουλειά εδώ και το ΕΛΚΑ θα στηρίξει ε, τις περισσότερες, έτσι, τις περισσότερες τροπολογίες στις συμβιβαστικές. Αυτά λέει η κυρία Βίρκουνεν. Και όπως βλέπετε βελτιώνεται και τα αγγλικά μου. Your English is, very good. Ναι, ναι, είναι πολύ καλά τα αγγλικά σας. Ε. Κύριε Ντεμεσμάκερ από την ομάδα ECR, έχετε το λόγο. Εγώ, Βίμ, πάλι θα μιλήσω Ολλανδικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια την κυρία Ταπαρντέλ και τους ε, συναδέλφου ε, για τις συμβαστικέ ε, τροπολογίες. Χαίρομαι που λάβατε υπόψη και τις δικές μας τροπολογίες και τις συμπεριλάβατε στην συμβαστική πρόταση. Οι τροπολογίε, κατά τη γνώμη μου, αντανακλούν τη σωστή ισορροπία. Οπότε από την δική μα πλευρά έχετε κάθε στήριξη. Οι συμβαστικές τροπολογίες διασφαλίζουν μια σωστή ε, προστασία των χρηστών και με την απαραίτητη ευελιξία για τις ε, διαδικτυακές πλατφόρμες. Είναι μια σημαντική πρόκληση σε αυτό το θέμα. Μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερη προστασία των ε, χρηστών. Για να έχουμε καλύτερη ισορροπία και σχέση μεταξύ αυτών των χρηστών και της διαδικτυακής πλατφόρμας. Και ο περιορισμός ε, της ρήτρα ε, ποιότητας ή του πλέον ευνοημένου πελάτη είναι μια θετική εξέλιξη. Διασφαλίζει ε, επιχειρηματική ελευθερία για τους επαγγελματίες χρήστες ή εμπορικούς χρήστες και προστασία του καταναλωτή από την άλλη, που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Μια σειρά χώρε έχουν ήδη δώσει ε, θετικό παράδειγμα, αλλά πρέπει να υπάρξει και ευρωπαϊκή προσέγγιση. Τέλος, είμαι πεπισμένο ότι με την προστασία του εμπορικού απορρίτου και άλλων ευαίσθητων πληροφοριών που ε, θα παρέχουν οι διεκτικές πλατφόρμες ε, είναι μια θετική εξέλιξη για να ε, προχωρήσουν περαιτέρω. Σας ευχαριστώ και πάλι. Νομίζω ότι αυτές οι τροπολογίες ανοίγουν τον δρόμο για, μια πιο, για ένα πιο δίκαιο ανταγωνισμό στο Ευρωπαϊκό Διαδίκτυο. Στο μάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τέλη της της ΑΛΤ. Ευχαριστώ κύριε Κόχα. Ευχαριστώ, Κλάουντια. Καταρχάς, θέλω να πω ότι στην Άλντε πιστεύουμε ότι είναι καλή νομοθετική πρόταση της Κομισιόν για τη δημιουργία ενός πλαισίου αλληλεπίδρασης των επιχειρηματικών χρηστών και των πλατφορμών. Εμείς ακολουθήσαμε στις διαβουλεύσεις στην ε, προσέγγιση του ότι απαιτείται βελτίωση σε κάποια στιγμή. Ίσως να τονίσει υπερβολικά μία πτυχή. Η Deutsche Bahn ε, κύριε ε, πουλάγανε πιστήρια πριν να υπάρξουν πλατφόρμες αυτές. Αλλά έχουμε όμως αυτήν την έλευση των πλατφορμών που δίνει ε, νέα στοιχεία. Ε, συγκρίσεις, νέες ευκαιρίες, προσφορές. Και σίγουρα όλα αυτά συνοδεύονται από νέες δυνατότητες και για τους επιχειρηματικούς χρήστες. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε την ουσία της νομοθεσίας. Απλά θέλουμε να βελτιώσουμε την πρόταση της Κομισιόν. Και με τις ευαισθητικές τροπολογίες καταφέραμε να τελειοποιήσουμε κάποιες πτυχές. Καλή πρόταση Κομισιόν, όπως είπαμε απλά. Νομίζω ότι την πήγαμε λίγο πιο μακριά εμείς. Οπότε θα πρότεινα να γίνουν δεκτές οι τροπολογίες, οι συμβαστικέ πλην μια μορισμό του κόστου στη διάρκεια της διαμεσολάβησης, το ξέρει και η συγκητρία. Αλλά σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, Νομίζω ότι είναι καλή η πρότασή μας από την ποιότητα της Κομισιόν και θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια. Σας ευχαριστούμε κύριε Τέλιτσκα. Κυρία Κίλενεν, Μύρια, για την ΚΟΕ. Thank you. Thank you, Mr. Koch, our chair. Uh, I want to thank Claudia. It has been great cooperation and also... Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω την Κλάουδια και για τη συνεργασία ε, μαζί μου και με τους υπόλοιπους συναδέλφους. Ε, ήταν πολύ ευχάριστη. Ε, νομίζω πως έχουμε όντως ισορροπημένη έκθεση και με χαρά θα πω ότι μπορούμε να στηρίξουμε αυτήν όλη τη δουλειά που έκανες. Δεν είναι συνηθισμένο να στηρίζουμε όλες τις τροπολογίες, αλλά αυτή τη φορά ναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Έκλεισε ο κατάλογος των σκιωδών εισηγητών. Ποια άλλη έχουν στήσει το λόγο. Κύριε Άντερσον, Λούση. Um, Ευχαριστώ. Ε, και εγώ θέλω να πω θετικά λόγια για τη δουλειά της εισηγήτριας ε, και είναι θετικό και νομικά και ε, αυτό που κάνει αυτή η έκθεση και σωστά είναι να προσθέσει περισσότερες λεπτομέρειες σε ένα θέμα που θα ήταν πολύ δύσκολο να επιβληθεί σύμφωνα με τον γενική ε, νομοθεσία περί ανταγωνισμού της Ένωσης που δεν είναι πάντοτε η κατάλληλα φτιαγμένη. Είναι πολύ χρήσιμο λοιπόν που εμείς συντάσσουμε έκθεση από αυτού, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα και όλοι μας θα έχουμε κάποιοι υπόψη μας, όπου οι μικρές ε, εταιρείε βασίζονται σε αυτού του είδους τις υπηρεσίες ε, και επηρεάζονται αρνητικά και άδικα από τα μεγάλα τέρατα, για να τα πω έτσι. Ε, μόνο λίγοι παρέχουν ε, τις μηχανές αναζήτησης ε, και γι' αυτό σας λέω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένη με αυτή τη δουλειά που κάναμε εδώ και εγώ και οι υπόλοιποι θα πρέπει να το προθέσουμε και στις άλλες επιτροπές. Ελπίζω και υπάρχουν κάποιες τροπολογίες που ψηφίζονται χωριστά ε, για τεχνικούς λόγους, αλλά τις οποίες ελπίζω πως θα μπορέσουμε να τις στηρίξουμε. Ε, ακούγονται τεχνικές, αλλά είναι σημαντικές για τις βοηθητικές ας πούμε, υπηρεσίες που δίνουν περισσότερη προστασία. Και να πω επίσης ότι πιστεύω πως είναι πολύ θετικό που έχουμε μια ρήτρα εδώ που αφορά τις μικρότερες ε, επιγραμμικές εταιρείε μπορούν σε αυτό να βασιστούν, γιατί θέλουμε αυτός ο κανονισμός να είναι ιδιαίτερα ε, ε, για τις μικρές ε, εταιρείε που ε, λειτουργούν επιγραμμικά. Ευχαριστώ και θα ελπίζω να υπερψηφιστεί και στην Ολομέλεια. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ τη Σάντρεσον Μας μένει η Κομισιόν. Να μας πείτε αν θεωρείτε και εσείς ότι έχουμε βελτιώσει την πρότασή σας. Ε. Ναι, γεια σας. Μιχαήλ Κιόνιγκ από τη Γάμα Δελτα Γκρό. Θέλω να σας ευχαριστήσω πράγματι για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις ε, και την συνεισφορά σας. Φυσικά και είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε βελτίωση που μπορεί να προσθεθεί σε μια πολύ καλή ήδη, όπως πιστεύουμε, πρόταση ιδίως αν παραμείνει αρχιτεκτονική και η έμφαση δοθεί ε, στη μεγαλύτερη διαφάνεια ίσως σε άλλους τομείς, ε, όπως αυτή που αναφέρατε για τους πρόστους διάβλους, το αντιλίστην κτλ. Εκεί συμφωνούμε με τη γενική φιλοσοφία της πρότασης. Εκεί που μπορεί να είμαστε λίγο πιο διστακτικοί είναι το να πάμε πολύ μακριά είναι μια προσέγγιση με δύο βήματα, σε ένα τομέα που αναπτύσσεται με ταχύς Το δεύτερο βήμα έχει ήδη δρομολογηθεί. Βλέπουμε την οικονομία αυτή των πλατφορμών και είμαστε λίγο πιο ε, επιφυλακτικοί σε ό,τι αφορά συγκεκριμένε πρακτικέ ή απαγορεύσει ή το οτιδήποτε έχει να κάνει με τι τιμέ, ε, τα τέλη, γιατί όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, είναι οριζόντιο μέτρο. Θα πρέπει λοιπόν να μπορεί να καλύψει όλες τις πλατφόρμες και όλους τους τομείς. Είμαστε όμως πεπισμένοι και αισιόδοξοι ότι μπορούμε να προχωρήσουμε γιατί και οι άλλες επιτροπές εργάζονται πάνω σε αυτή την πολύ σημαντική αυτή πρόταση και έχουμε προχωρήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κένιχ. Ένα άλλο όνομα είχα μπροστά μου εγώ, αλλά δεν πειράζει. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρατήρησή σας. Και τώρα θα δώσω ξανά το λόγο στην εισηγήτρια για να κλείσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω ακόμη μια φορά τους συναδέλφους, σκιώδεις εισηγητές,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 να ευχαριστήσω τον Λούκας Μικέλγα και τους ε, συναδέλφους του, της, της γραμματείας της Επιτροπής που με βοήθησαν πολύ. Προσπάθησα στην ε, ε, έκθεση αυτή να έχω μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για να αποφύγουμε τον κατακαρματισμό που υπάρχει στα, ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Μιλάμε για την ψηφιακή αγορά που προχωράει και εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα και εμείς τρέχουμε για να προλάβουμε τις εξελίξεις στην αγορά αυτή. Οφείλουμε λοιπόν εμείς ως Ευρωπαίοι νομοθέτες να ε, επιφέρουμε μια ισορροπία στην αγορά αυτή, ισορροπία ανάμεσα στην ε, ψηφιακή αγορά και την παραδοσιακή αγορά. Αυτή η ισορροπία λοιπόν θα πρέπει να βρεθεί για χάρη των ε, τελικών χρηστών και καταναλωτών. Νομίζω πως εδώ αυτό το καταφέραμε. Είναι μια έκθεση που βασίζεται στην πρόταση της Κομισιόν, που αγγίζει όλους τους τομείς δραστηριότητα, αλλά όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, όταν βλέπουμε αυτές τις πλατφόρμες ε, ε, που λειτουργούν online, κυρίως αφορούν τον τουρισμό και τις μεταφορές. Και έχουμε πολλές εταιρείες που εργάζονται μέσω των επιγραμμικών ε, πλατφορμών και γι' αυτό και θα πρέπει εμείς να έχουμε σαφή, ε, μια σαφή ε, και διαφανή νομοθεσία που θα επιτρέψει σε αυτές τις εταιρείες να λειτουργήσουν ομαλά προς όφελος των προμηθευτών και των καταναλωτών. Ευχαριστώ ακόμα μια φορά για αυτή τη συνεργασία και ελπίζω πως αυτή η γνωμοδότηση θα χρησιμεύσει και στους συναδέλφους της ΣΥΜΚΟ. Ευχαριστούμε πολύ την Πέμπτη ε, αύριο 22 θα ψηφίσουμε και προχωρούμε στο σημείο 7 που είναι πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Κλάντια Σμίτα Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι έχουμε μπροστά μας ένα τεχνικό θέμα που δεν ε, είναι τόσο επίμαχο με, όπως άλλα θέματα, όπως παραδείγματο χάρη αυτό με τη κινητικότητα. Ε, ε, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι μια καλή αφετηρία. Έχουμε συναντήσεις με τους σκιοδησηγητές και νομίζω ότι αυτό το οποίο ε, προέκυψε μέχρι τώρα είναι ότι θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα πιο πέρα από την πρόταση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που θα είναι στραμμένο προς το μέλλον και που θα λαμβάνει υπόψη κάτι πάρα πολύ αναγκαίο που είναι η πρόθεση της ψηφιοποίησης. Αν εφαρμοστεί αυτή η έκθεση ε, θα έχει καλύτερα ε, πρότυπα, θα μειωθούν οι τιμές, θα υπάρξει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τις πληροφορίες για τις ηλεκτρονικές εμπορευματικές ε, μεταφορές, έχουμε και τη βιομηχανία 4.0. 20 εκατομμύρια ε, εργατόρες ε, πώς ε, δαπανώνται. Δαπανώνται γιατί πρέπει να μεταφέρονται στον υπολογιστή τα δεδομένα, να εκτυπώνονται και ξανά τα ίδια και μπορεί να γίνεται πέντε φορές ανα αποστολή το ίδιο πράγμα. Και νομίζω ότι αυτό σημαίνει τεράστια καθυστέρηση και σπατάλη χρόνου και είναι και παράλογο Επίσης θα πρέπει να υπάρξει τυποποίηση της ε, κοινοποίηση ε, ε, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες. Πιστεύω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας εδώ τις πολυτροπικές μεταφορές και να κάνουμε κάθε προσπάθεια ώστε τουλάχιστον η ανταλλαγή πληροφοριών να γίνεται πιο, ως το δυνατόν πιο ομαλά και αποτελεσματικά. Σίγουρα είδαμε το 2018 ότι το 99% ε, των σφαλμάτων θα μπορούσαν να αποφευχθούν, αν μπορούμε να είμαστε ακόμα πιο αποτελεσματικοί. Και νομίζω ότι θα μπορούσε αυτή η έκθεση να δημιουργήσει ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο. Για τις αρμόδιες αρχές θέλω να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια ε, η οποία λαμβάνει υπόψη τις δικές μας απόψεις και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια πρόταση που θα βρει σύμφωνη την πλειοψηφία. Ε, θα πρέπει επίσης ε, η ε, αστυνομία να βλέπει τα εκτυπωμένα έγγραφα κάθε φορά, παραδείγματος χάρη τις φορτωτικές των φορτηγών και αυτό δίνει, καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί καθυστερήσεις και ιδίως λαμβάνοντας υπόψη την αυτοματοποίηση, μηχανοργάνωση και την ψηφιοποίηση που όλο και περισσότερο εξελιστεί. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα τα οποία μπορούμε να βελτιώσουμε. Το πρώτο βήμα είναι να υπάρχει η, ηλεκτρονική, η αποδοχή των ηλεκτρονικών ε, αιτήσεων και άλλων εγγράφων από τις αρχές. Εδώ μιλάμε βέβαια για το 2020-2025 ε, ε, υποχρεωτική ηλεκτρονική διαβίβαση των δεδομένων. Πρέπει να πω ότι έχω έρθει σε επαφή με πολλούς ε, εκπροσώπους του κλάδου των μεταφορών, ε, ε, της επιβολής του νόμου, εκπροσώπους αστυνομίας κτλ. κτλ. Σίγουρα υπάρχουν ακόμη κάποια ανοιχτά σημεία τα οποία θα τα συζητήσουμε. Δεν πιστεύω ότι οι θέσει εργασίας ε, ε, που απαιτούνται ε, για να υπάρχουν αυτές 120 εκατομμύρια εργατόρες ότι θα καταργηθούν όλες αυτές δεν νομίζω ότι περί αυτού πρόκειται ελπίζω ότι με τη συνεργασία μας με το Σκιώδη θα συνεχίσουμε να προχωρούμε και θα βρούμε το σωστό μείγμα και της ενίσχυσης αλλά και των απαιτήσεων που πρέπει να υπάρχουν ώστε η οικονομία, η συνεργασία και οι συναλλαγές με τη διοίκηση να βελτιωθούν και όλη αυτή η γραφειοκρατία, η αχρίαστη, να μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ευχαριστώ πολύ, Κλάουντια λέει ο πρόεδρο, και περνάμε στου κοιόδε εισηγητέ για την ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Ζαμπέλ Ντεμόντε. Ε, ευχαριστώ. Καταρχάς να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Κλάουδια Σμίτ για την εργασία που έχει κάνει και επειδή ανάμειξε όλα τα μέρη στην επεξεργασία αυτής της έκθεσης. Ε, όλα είναι και πιο ψηφιακή γίνεται η εποχή μας και πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες για να προσαρμοστούμε στις αλλαγές και στον τομέα των μεταφορών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και μπορεί να οδηγήσει σε απλοποιήσεις ε, και σε μια ελάφρυνση των διαδικασιών, κυρίως εκείνης της διαδικασίας ελέγχου. Πιστεύω πως αυτό θα πρέπει να συμβαδίσει με την εξέλιξη του ψηφιακού ταχογράφου ε, ταχυγράφου που θα πρέπει να μπορεί να αποθηκεύει όλες τις πληροφορίες ανεξάρτητα από το ποια θα είναι τα αποτελέσματα του ε, πακέτου για την κινητικότητα πιστεύω πως το περιεχόμενο αυτού του φακέλου θα πρέπει να είναι παρόμοιο ή εν πάση περιπτώσει συνεχτικό ε, με το θέμα. Όσον αφορά τις ε, πληροφορίες που ανταλλάσσονται και τα δεδομένα θα πρέπει αυτά να τα διαχειρίζεται ένα κεντρικό σημείο. Δεν θα είναι εύκολο αλλά θα πρέπει ωστόσο να είναι εναρμονισμένες. Η πρόταση αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει λύση για την αντιμετώπιση της έλλειψης ε, ομοιόμορφων εγγράφων εγγράφων ε, αλλά θα βοηθήσει και στις ε, αρχές της τάξης να ε, βελτιώσουν και να απλοποιήσουν τις διαδικασίες, αλλά και να τις ε, κάνουν και εξ αποστάσεως, χωρίς να χρειάζεται να σταματήσουν δηλαδή το φορτηγό. Κέρδος χρόνου και αποτελεσματικότητας λοιπόν στους ελέγχους, τόσο για τους οδηγούς είναι αυτό ωφέλιμο, όσο και για τις δυνάμεις τις αστυνομικές. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα διεθνή πρότυπα όταν αποφασίζουμε να φτιάξουμε ένα ευρωπαϊκό πρότυπο για τα ηλεκτρονικά έγγραφα μεταφορών, ώστε να μην υπάρχουν διαφορές στο μέλλον ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ένωσης και τα τρίτα κράτη. Και τέλος θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τη δυνατότητα τροπολογίας για να αντιμετωπίσω και άλλο ένα σημείο που είναι πολύ σημαντικό για μένα που είναι η προστασία των ζώων των ζώων γιατί και ως προς αυτό δυστυχώς υπάρχουν καταχρήσεις οι οποίες θα πρέπει να αποφευχθούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ντεμόντε. Από το Εκείς ε, είσαστε εδώ κύριε Ζλωτόφσκι, παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Σμιτ ε, για το έργο της. Η ομάδα μας στηρίζει πλήρως οποιαδήποτε πρωτοβουλία που θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη ψηφιοποίηση τομέα των ε, μεταφορών όπως ε, η διαβίωση των δεδομένων για παράδειγμα, ηλεκτρονικές επικοινωνίες μεταξύ των μεταφορικών εταιριών και των αρχών των κρατών μελών ε, είναι κάτι αναγκαίο κατά εμάς για τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη μείωση του κόστους και είναι κρίμα που δεν εντάσσεται στο σχέδιο της κινητικότητας το λόγο έγγραφο θα μπορούσε πιστεύω να μπει ε, στο σκέλος που έχει να κάνει με την εφαρμογή της νομοθεσίας και την ε, οικονομία της αγοράς. Σε ό,τι αφορά την πρόταση 26, σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή οδηγία, νομίζω ότι εδώ είναι λίγο υπερβολικό αυτό που προτείνεται. Όσο δεν λειτουργεί αυτό το σύστημα ακόμη, δεν νομίζω ότι αιτιολογείται κάτι τέτοιο ε, και δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε ε, ακόμη το πόσο καλά ε, θα είναι τα αποτελέσματα αυτού του συστήματος. Σε ό,τι διάφορα την χρήση και τη συγκέντρωση αυτών των ε, στοιχείων ε, θα ήταν κάτι θετικό, ε, αλλά πρέπει να υπάρχει μια μεταβατική περίοδος σε ό,τι αφορά την τροπολογία 17 για να περάσουμε δηλαδή από, τις, το χαρτί, τις έντυπες αυτές δηλώσεις στις ηλεκτρονικές Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις ομεκασίες επιχειρήσεις. Το άρθρο 15 πρέπει να λάβει υπόψη τις ιδιαιτερότητες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτή την αναθεώρηση μετά από πέντε χρόνια. Δεν αρκεί να λέμε δύο χρόνια, δεν είναι επαρκής η περίοδος αυτή. Θα κάνουμε και συγκεκριμένε προτάσεις και προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία μας με την ΣΥΤΑ και τους Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος, κ. Λωτός και περνάμε στην Άλντε. Κυρία Μπιλμπάου, Μπιλμπάου Μπαραντίκα. Καλημέρα σας σε όλους και όλες. Καταρχά να ευχαριστήσω ε, την εισηγήτρια για την εργασία που έκανε και για τη διάθεση που έδειξε απέναντι σε όλες τις ε, ομάδες των εργαζομένων στα γραφεία. Ε, ήταν πραγματικά πολύ ανοιχτή για να πετύχουμε συμφωνία σε μια τόσο σημαντική έκθεση. Να πω Καταρχάς, ποιος είναι ο γενικός στόχος αυτής της έκθεσης, το να μπορέσουμε να καταφέρουμε ε, η βιομηχανία μεταφορών της Ευρώπης να έχει ηγετικό ρόλο στην εναρμόνιση και στην... Ε, έχουμε κουραστεί να τα βλέπουμε όλα αυτά. Η μεταφορά προϊόντων, εμπορευμάτων αυξάνεται διαρκώς και θα συνεχιστεί η αύξηση αυτή και στα επόμενα χρόνια. Τι συμβαίνει το 99% των γράφων που ε, φορτωτικών στις διασυνοριακές ε, μεταφορές ε, χρησιμοποιεί το χαρτί και το να μπορέσουμε να έχουμε σε ηλεκτρονική μορφή όλο αυτό το χαρτί ε, αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες. αυτό και πρώτο και κύριο γιατί οι αρχές δεν κάνουν τις κατάλληλη προσπάθεια που πρέπει να γίνει ε, να, να καταργηθεί το χαρτί και να μετατραπούν όλα αυτά σε ηλεκτρονική μορφή. Άρα λοιπόν πρέπει να λύσουμε δύο βασικά προβλήματα γιατί δεν έχουμε ένα πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε ένα πλαίσιο με διαφορετικά συστήματα ε, πολύ κατακαιρματισμένα που πρέπει να τα εναρμονίσουμε και έπειτα έχουμε και συστήματα τα οποία δεν είναι διαλειτουργικά. Αυτή είναι η μαγική λέξη για ένα σωρό εκθέσεις στις μεταφορές. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα διαλειτουργικό ανάμεσα στα κράτη και ανάμεσα στις πλατφόρμες των διαφόρων ε, επιχειρήσεων. Το θέμα είναι πώς θα το λύσουμε λοιπόν αυτό το θέμα. Άλλη μαγική λέξη είναι η συνοχή σε όλες αυτές τις εκθέσεις για τις οποίες μιλάμε. Αυτή η έκθεση είναι κομμάτι ε, της στρατηγικής κινητικότητας ε, Ευρώπης σε κίνηση. Τι, τι θέλουμε να κάνουμε, το ίδιο, να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε την διαλειτουργικότητα Άρα λοιπόν και εδώ το ίδιο και γι' αυτό και εκτιμώ θετικά τις τροπολογίες που υπέβαλε η εισηγήτρια. και την τροπολογία 3 που μιλά για συνοχή στο ψήφισμα και συνοχή με την έκθεση του 17 όπου καλεί τα κράτη να δέχονται ηλεκτρονικά έγγραφα στις εμπορευματικές μεταφορές και να χρησιμοποιηθεί το σύστημα CMR χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση. Γι' αυτό θεωρούμε πως οι αρχές θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές να ξεκινήσουν και να αναπτύξουν τους απαραίτητους μηχανισμούς ώστε να μπορούν να λαμβάνουν τις πληροφορίες με ηλεκτρονικό τρόπο. Δεν μπορούμε εδώ πια να δείξουμε άλλη ελαστικότητα, πρέπει να το κάνουν. Και οι οικονομικοί φορείς επίσης θα πρέπει να αρχίσουν να χρησιμοποιούν αυτό, να ετοιμάζονται για να χρησιμοποιήσουν αυτού του είδους τις ηλεκτρονικές, τα ηλεκτρονικά έγγραφα. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, στην ουσία ε, βλάπτουμε τις μικρομεσαίες αλλά και τις μεγάλες εταιρείες που ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν μηχανισμούς για να είναι πιο αποτελεσματικές ως εταιρείε, για να καταργήσουν το χαρτί, για να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και μεγαλύτερη ταχύτητα ε, στις ε, μεταφορές. Γι' αυτό και πιστεύω πως είναι απαραίτητη μια τυποποίηση των πληροφοριών που είναι απαραίτητες ώστε όλοι να μπορούμε να αναπτύξουμε αυτό το σύστημα ε, εναρμονισμένα. Χρειάζεται λοιπόν, χρειάζονται στάνταρ, πρότυπα, κοινέ διαδικασίες και μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να εξαλείψουμε αυτά τα προβλήματα που έχουμε τώρα λόγω της του κατακαιρματισμού και της μη διαλειτουργικότητας των συστημάτων. Και σε αυτή τη γραμμή θα είναι και οι τροπολογίες μας αυτές ε, τις οποίες δουλεύουμε με την κυρία Εσμύρ και ελπίζουμε πως θα μπορέσουμε να έχουμε ε, ε, την κυρία Σμιθ και να δούμε και να έχουμε έτσι ένα ε, ομοιόμορφο, όπως είπα, σύστημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μπιλμπάο. Η κυρία... Thanks to η κυρία Κιλώνεν από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ πολύ την Κλάοντια και ε, να πω ότι ήδη έχουμε κάνει πολύ θετικές ε, συζητήσεις ε, και ειδικά για το ε, σύνταξη του σχεδίου έκθεσης ε, μου άρεσε πολύ αυτή η πρόταση ότι η Κομισιόν θα πρέπει αμέσως να ξεκινήσει την εργασία της επί των απαραίτητων κατεξοδότηση πράξεων για να αποφύγουμε περαιτέρω καθυστερήσεις. Πάρα πολύ χρόνο έχουμε φάει με αυτό το πακέτο κινητικότητας. Και Χρειαζόμαστε κατεπηγόντως το σύστημα της κοινή πλατφόρμας ώστε να μπορούμε να μοιραζόμαστε έγκαιρα ε, και σε πραγματικό χρόνο αυτές τις πληροφορίες. Ελπίζω λοιπόν ότι θα προχωρήσουμε πιο γρήγορα από ό,τι στο παρελθόν και θα εξοικονομήσουμε και το σημερινό μας χρόνο. Γι' αυτό σταματώ αμέσως. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ καλή δουλειά κάνετε και θα συνεχίσουμε μαζί να βρει, στην αναζήτηση ακόμη καλύτερων λύσεων. Μπορούμε μαζί να τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Μύρια. Δεν βλέπω να θέλει το λόγο κάποιο εκπρόσωπο κάποια άλλη πολιτική ομάδα. Οπότε πηγαίνουμε ευθύ αμέσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σάντρο Σανταμάτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Αρχικά, να εκφράσω τις ευχαριστίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τον εισηγητή και όσους συνέβαλαν ε, σε αυτό το έργο και την σαφή στήριξη προς αυτή την πρωτοβουλία που αντανακλάται και στο σχέδιο έκθεσης. Είναι πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία. Μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση σημαντικού διοικητικού κόστους από πλευράς ε, των ε, εμπορευομένων και είναι και σημαντικό βήμα στην, προς την ψηφιοποίηση του κλάδου και ένα σημαντικό βήμα προς την ε, εναρμόνιση σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταφορών το οποίο ανέφεραν ορισμένοι στις παρεμβάσεις τους. Κάτι το οποίο θεωρούμε πράγματι σημαντικό. Μία εναρμόνιση που και εμείς θεωρούμε και επιβεβαιώνουμε ότι θα συνάδει με τα διεθνή πρότυπα. Είδαμε ότι η πρόταση ε, υποβάλλει μία προσέγγιση που είναι ακόμα πιο φιλόδοξη σε σχέση με αυτή που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ιδίω ε, σε ό,τι αφορά την υποχρεωτική διάσταση του συστήματος για όλους τους χρήστες και επέκταση ε, του πεδίου εφαρμογής και σε άλλε μορφές εγγράφων. Αυτό που είχε εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, ε, τα είχαμε εξετάσει τέλο πάντων όλα αυτά πριν υποβάλουμε την πρόταση και καταλήξαμε στο συμπέρασμα τουλάχιστον στην αρχή παρότι η δική σας έκθεση μπορεί να προκαταλαμβάνει ορισμένες μελλοντικές εξελίξεις, θα προτιμούσαμε ένα υποχρεωτικό σύστημα ε, που θα είναι υποχρεωτικό για τις αρχές, αλλά προαιρετικό για τον ε, εμπορευόμενο. Έως ότου οι υπηρεσίες που είναι απαραίτητες και συνδέονται με τα ψηφιακά έγγραφα θα έχουν αναπτυχθεί επαρκώς και τότε το κόστος ε, θα είναι πολύ χαμηλό. Επομένω, ε, στην αρχή προτιμούμε να δώσουμε τη ε, δυνατότητα στους εμπορευμένου να επιλέξουν αν θέλουν να αξιοποιήσουν ψηφιακέ πληροφορίες ή να συνεχίσουν τις συνήθεις πρακτικές. Αλλά είμαστε πεπισμένοι ότι πολύ σύντομα όλοι θα δουν ε, το πλεονέκτημα της χρήσης ψηφιακών πληροφοριών. Σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή χρήση αυτού του συστήματος και σε άλλες μορφές εγγράφων, πρέπει εδώ να γίνει μια διάκριση μεταξύ πληροφοριών ε, των επιχειρήσεων προς την κυβέρνηση, πληροφοριών που είναι μεταξύ κυβερνήσεων και πληροφοριών που είναι μεταξύ επιχειρήσεων. Συμφωνούμε λοιπόν ότι είναι σημαντικό να υπάρχει διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων. Όμως, από την άλλη, θα πρέπει να βρούμε και την πλέον κατάλληλη προσέγγιση σε αυτές τις διαφορετικές μορφές ε, επικοινωνίας. Γι' αυτό και στην πρόταση λέγαμε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε ε, αρχικά εφαρμόζοντας την πρόταση στις πληροφορίες των επιχειρήσεων προς τις κυβερνήσεις. Σας ευχαριστώ και πάλι για τη στήριξη. Βλέπω ότι συμμερίζεστε κι εσείς τη γνώμη μας ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η πρόταση και σας ευχαριστούμε και εμεί ευχαριστούμε κύριε Σανταμάτο. Ό,τι βοηθάει στη μέση τη γραφειοκρατία, μας βρίσκει εμά ε, το κοινούλιο στο πλευρό σα. Για να κλείσει η κυρία Κλόντια Σμιτ. Με τι 11 έχεις. Μία και μόνη ευκαιρία. Είναι η ευκαιρία σου. Ναι. Εντάξει, να μην ε, κρατήσει και τόσο. Φυσικά ε, πρέπει να πω ότι πήραμε την άποψη πολλών αρχών και επιχειρήσεων και στο θέμα των ελέγχων θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με την ψηφιοποίηση στα, στα φορτηγά ε, μήπως μπορεί να οι έλεγχοι ε, που δεν θα είναι πλέον φυσικοί ε, να δημιουργήσουν πρόβλημα όταν μεταφέρονται παραδείγματος χάρη απλά μετανάστες ή οτιδήποτε. σίγουρα θέλουμε να δώσουμε μια όθηση προς τη σωστή κατεύθυνση για να πετύχουμε κάποια πράγματα και πρέπει και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ακολουθήσουν. Δεν μπορούμε όμως να περιμένουμε 30 χρόνια για να συμφωνήσουν ότι θα ακολουθήσουν οι ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, πρέπει ήδη από τώρα ε, να κερδίσουμε κάποιο χρόνο και να προχωρήσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά για μια ακόμη φορά τους συναδέλφους από τις άλλες πολιτικές ομάδες ήταν η πρώτη έκθεση που από την αρχή τόσο ανοιχτό πνεύμα επικράτησε. Μιλήσαμε όλοι ε, πάρα πολύ ανοιχτά, ειλικρινά και όλοι είμαστε στην ίδια γραμμή. Και ελπίζω και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δεχθεί ως είναι αυτή η πρόταση, δηλαδή να βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Σε ό,τι αφορά την προθεσμία αποβολής ε, τροπολογιών 4 ε, Δεκεμβρίου 10 το πρωί. Οπότε όλοι μπορείτε να τοποθετηθείτε και τώρα μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 8. Δεν είναι όμως εδώ ο εισηγητής. Γιατί προβλεπόταν στις 11. Οπότε προβλέπω, ε, προτείνω συγγνώμη να κάνουμε ένα δεκάλεπτο διάλειμμα. So, wir setzen unsere Beratung fort. Ich hoffe, dass alle wieder da Τέλειωσαν ε, οι διαβουλεύσεις ε, ή το διάλειμμα για καφέ. Περνάμε λοιπόν στο επόμενο σημείο της ημερήσια διάταξης ε, για την πρόταση κανονισμού σε ό,τι αφορά το κανονισμό του 2009 για ένα κώδικα θεώρησης διαβατηρίων. Η Ορχέλη είναι ο εισηγητής μας. Α, εκεί στην άκρη. Παρακαλώ. Έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι. Στον τομέα του τουρισμού και των μεταφορών ήδη έχουμε καταλήξει σε πολλά συμπεράσματα σε ό,τι αφορά το προηγούμενο πακέτο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι θεωρήσει για τον κώδικα θεωρήσεων και τουριστική θεώρηση πριν από τρία χρόνια, αν θυμάστε. Η νέα πρόταση της Κομισιόν έχει ως στόχο να απλοποιήσει τις ε, διαδικασίες για τις ε, μικρές διάρκειας θεωρήσεις ε, τι τουριστικές. Υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ διαφόρων πτυχών για να φέρνουμε περισσότερους τουρίστες στον χώρο Ζένγκεν μέσω μέτρων διευκόλυνσης, χωρίς όμως να διακινδυνεύουμε την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. Έτσι θα υπάρχει και αύξηση στον τομέα του τουρισμού και των μεταφορών και νέες θέσεις απασχόλησης. Έτσι η Ευρώπη θα γίνει ε, υπαριθμόν ένα τουριστικό προορισμός. Η πρόταση απλοποιεί ε, τις διαδικασίες για όσους θέλουν να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μικρή διάρκεια ε, παραμονή. Ε, εξοικονομούν έτσι και χρήματα και διοικητικό άχθος. Η ψηφοφορία σε σχέση με την ψηφοφορία στην Ολομέλεια και με την πρώτη πρόταση, υπάρχουν κάποια στοιχεία που δεν υπάρχουν στην νέα πρόταση Κομισιόν. Το υποχρεωτικό θέμα των, πολλα... των θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων έχει αλλάξει. Για να μην έχουμε το σύστημα Cascade. Η έννοια της τουριστικής θεώρησης και η ιδέα των επαγγελματιών του αθλητισμού και του πολιτισμού επίση είναι κάτι το οποίο που λείπει. Αυτό δεν δείχνει μια θετική προσέγγιση προ το έτος ε, πολιτισμική κληρονομιά στην Ευρώπη. Τέλος, ε, δεν ε, εξηγείται γιατί αυξάνεται το κόστο ορισμένων θεωρήσεων. Εγώ επικεντρώθηκα στις εξής αρχές να αυξήσουμε την πιθανή περίοδο διάρκειας των θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων στα 10 έτη, έως τα 10 έτη, για, τους, ε, για συγκεκριμένους ε, ταξιδιώτες. Να διατηρήσουμε τη σημερινή διάταξη που αφορά μεγαλύτερη διάρκεια θεωρήσεων για τους MEVs, αντί για το σύστημα Cascade που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν θα αυξήσει την ε, ε, έκδοση των θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων. Η παρατεταμένη παραμονή στην ε, Ευρώπη έτσι θα διατηρείται για συγκεκριμένους ταξιδιώτες. Να επιμένουμε στους ετούντε να υποβάλουν αίτηση σε προξενείο άλλου κρατούς μέλους όταν το προξενείο του οικίου και τους απέχει πάνω από 500 χιλιόμετρα από την ε, διαμονή τους. Ιδίω σε μεγάλες χώρες όπως η ε, Ινδία, η Κίνα, αυτό είναι σημαντικό πρόβλημα. Ένα ποσοστό του αυξημένου τέλους να διοχετευτεί για τη στήριξη της κοινή ε, προαγωγής της τουριστικής στρατηγικής. Υπάρχουν εξαιρετικά παραδείγματα γι' αυτό και γι' αυτό θα θέλαμε να συμπεριληφθεί στον κώδικα θεωρήσεων. 85 τροπολογίες είχαμε συνολικά. Έχω καταρτήσει 5 συμβαστικές τροπολογίες που θα συζητήσουμε απόψε στη συνάντηση των σκιωδών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές και τους συναδέλφους. Και ελπίζω να έχουμε έναν καλύτερο κώδικα θεωρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. <laughs> Σε ευχαριστώ. Τέλεια το είπατε στα Ουγγρικά, Πρόεδρε. Περνάμε στου σκιώδεις συζητητές από το ΕΛΚΑ. Κυρία Κλούν. Δίρντρε. Thank you. Thank you very much, Chairman. And, uh, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ ε, που μου δίνετε το λόγο στη θέση του Κλάουδιο Μοντενέρο που δεν μπορούσε να είναι σήμερα εδώ. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή Ιστβαν για την παρουσίαση της γνωμοδότησης που αγγίζει σημαντικά θέματα για τη διευκόλυνση των διαδικασιών έκδοσης θεωρήσεων. Ε, η πρόταση της Κομισιόν αντικατοπτρίζει κάποια σημεία κλειδιά που ήδη συζητήθηκαν στην προηγούμενη ε, αναθεώρηση του 2014 και που λόγω των αποκλεινουσών απόψεων δεν προχώρησε. Ας μην ξεχάσουμε ε, ότι ο ευρωπαϊκός προορισμός είναι από τους πιο περιοριστικούς όσον αφορά τις απαιτήσεις ε, θεωρήσεων. Σύμφωνα με την έκθεση αυτό το άνοιγμα του 2018 από το Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού είμαστε πολύ κάτω του μέσου όρου για τη, όσον αφορά τη διευκόλυνση θεωρήσεων. Θέλω να υπογραμμίσω δύο σημεία. Η γνωμοδότηση θα πρέπει να εστιάζεται μόνο στη βελτίωση των κανόνων του κώδικα θεωρήσεων για τις ε, θεωρήσεις μικρής διάρκειας και έπειτα οι ετούντες που απορρίφθηκε το αίτημά τους θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα για έφεση και η δυνητική αποζημίωση θα πρέπει να προκύπτει από απόφαση δικαστηρίου και όχι ε, να απορρέει από αυτόν εδώ τον κανονισμό. Online πλατφόρμα λοιπόν για διαφανείς και αποτελεσματικές διαδικασίες έκδοσης θεωρήσεων. Η δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών ε, μέσων ε, χρειάζεται. Και όσον αφορά την ε, καταχώρηση του κόστος των θεωρήσεων για προώθηση τουριστικών δράσεων ε, αναγνωρίζω τη χρησιμότητα, ωστόσο από πρακτικής πλευράς το βλέπω δύσκολο. Το Κοινοβούλιο λοιπόν θα πρέπει να ολοκληρώσει αυτή την υπόθεση πριν από τις επόμενες εκλογές. Ευχαριστώ. Λυσία. Κύριε Σλοτόφσκι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κατά τη δική μας εκτίμηση πρόκειται για ένα πολύ καλό σχέδιο έκθεση το οποίο καλύπτει τα βασικότερα ζητήματα με τα οποία ε, απασχολούμαστε εδώ στην Επιτροπή μας. Ε, ο κώδικας θεωρήσεων λοιπόν είναι ε, μια πάρα πολύ καλή έκθεση αυτή, γι' αυτό και δεν καταθέσαμε καμία τροπολογία. πιστεύω ότι εμείς πρέπει να εστιάσουμε στη, στα δικής μας αρμοδιότητας ζητήματα, δηλαδή διαδικασίες απόξη θεώρησης για τις μεταφορές. και σίγουρα μπορούν να αξιοποιηθούν χρησιμοποιηθούν και τα ψηφιακά ε, μέσα για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων και την επαλήθευση των δεδομένων από 23 των χωρών. Ε, νομίζω ότι πάρα πολύ γρήγορα θα καταφέρουμε να ε, ολοκληρώσουμε το έργο πάνω σε αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος για την Άλντε. Εσείς κύριε Ράτας. Kao što η πρώτη συζήτηση ε, για αυτό τον ε, κώδικα και σε αυτή τη συνεδρία είχαμε πει ότι στηρίζουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και τις ε, βελτιώσεις που προτείνει ο εισηγητής. Είπαμε ότι θα καταθέσουμε τροπολογίες για την περαιτέρω απλούστευση της διαδικασίας και αυτό πράξαμε προκειμένου και να πετύχουμε μία αντίστοιχη, παρόμοια μάλλον, αν όχι ενιαία διαδικασία σε όλα τα κράτη-μέλη. Σε μια τροπολογία αναφέρεται και η διαθεσιμότητα της ψηφιακής έκδοσης ε, θεωρήσεων. Θα πρέπει να δίνεται και αυτή η δυνατότητα σε άτομα με αναπηρίες. Ε, να μένουμε και οι δικές μας προτάσεις να ληφθούν υπόψη στις συμβαστικές τροπολογίες, να υπάρξει καλή συνεργασία για να έχουμε τελικά μια καλύτερη δικασία έκδοση θεωρήσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και Ράντος. Γκουε. Με κύλωνε. Έχετε το λόγο. Ένα ευχαριστώ έχω This is not my, my... ευχαριστώ έχω μόνο να πω στον Ίστο. Δεν είμαι εγώ ευτυχώ ε, αρμόδια για όλα τα θέματα, άρα δεν είμαι υπεύθυνη για αυτή την έκθεση. Ιστβαν, ε, όμω έκανε πολύ καλή δουλειά, διάβασε και τι τροπολογίε σου. Και νομίζω ότι με καλή συνεργασία και η ΓΟΕ θα συνεισφέρει, θα βρούμε μια πολύ καλή λύση. Okay, Μάλιστα. Ε, ολοκληρώσαμε τον κύκλο των, τον γύρο των σκιωδών. Τον, ε, κυρία Ντεμόντ έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παίρνω το λόγο καταρχάς για να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική του πρόταση και με την ευκαιρία για να θυμίσω κάπως ε, το γενικότερο πλαίσιο αυτής της πρότασης κανονισμού γιατί αρχικά ο στόχος ήταν να περιοριστεί η ε, ε, παράνομη μετανάστευση και για διάφορους λόγους υπήρξε ε, μία πάυση των διαπραγματεύσεων εφόσον υπήρχε μία διαφορά ουσιαστική, δηλαδή να θεωρηθεί το άνοιγμα για αυτές τις θεωρήσεις ότι θα οδηγούσε σε αύξηση των τρομοκρατικών επιθέσεων. Αυτό θα πρέπει λοιπόν να ξεπεραστεί Αντίθετα, ε, πρέπει να διευκολύνουμε την πρόσβαση στον χώρο Σέγγεν για ανθρώπους που θέλουν να επισκεφθούν φίλους και συγγενείς ή για τα ε, επαγγελματικά ταξίδια, αλλά και το θέμα της προώθησης του τουρισμού είναι πολύ σημαντικό. Έγινε και μία μελέτη αντικτύπου ε, πρόσφατα και έδειχνε την τεράστιο αντίκτυπο Μάλιστα 150 δις ε, υποτίθεται ότι θα ε, προσφέρει η αύξηση η τουριστική στην επόμενη πενταετία και χάρη στις τουριστικές θεωρήσεις που δεν θα πρέπει να αποκλείονται. Συμμερίζομαι τις επικρίσεις λοιπόν που ασχέθηκαν σε αυτό το σημείο. Θα πρέπει λοιπόν να διευκολυθούν αυτές οι συμφωνίες για να, για να μην υπάρξουν εμπόδια στα κράτη-μέλη και επειδή είναι σαφές ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα ηλεκτρονικά συστήματα που υπάρχουν για την υποβολή των ετοιμάτων. Είμαστε στο σωστό δρόμο και ευχαριστώ και πάλι τον εισηγητή για την πρότασή του. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω να θέλει κάποιο άλλο το λόγο. Δεν ε, θέλει το λόγο ούτε η Κομισιόν, άρα να ξαναδώσω το λόγο στον Ιστβαν, τον εισηγητή μας. Ευχαριστώ ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα συναντήσω τους σκιώδεις σήμερα το απόγευμα και νομίζω ότι εκεί θα κλείσουν και όλα τα ζητήματα και θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Άτιλα, ένα μεγάλο ευχαριστώ, αλλά και να ευχαριστήσω και όλες τις άλλες ομάδες που μας στήριξαν. Ευχαριστώ πολύ. Τέσσερις το μεσημέρι στις 3 Δεκεμβρίου θα ψηφίσουμε για την έκθεση αυτή και τώρα πάμε στο τελευταίο σημείο της ε, δημόσιας συνεδρίασης ε, για ε, σήμερα που αφορά σχέδιο απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη εκ μέρου ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση τροποποίηση συμφωνία μεταξύ ΕΠΑ και Ευρωπαϊκή Κοινότητα όσον αφορά τη συνεργασία για την κανονιστική ρύθμιση τη ασφάλεια πολιτική αεροπορία. Κυρία Γκρίφιν δεν είναι εδώ. Κυρία Ουλσφκοφ θα την αντικαταστήσει. Σας ευχαριστώ, ναι πράγματι, προσωπώ την Τερέσα Γκρίφ που Λυπάται που δεν μπορεί να είναι πάρους. Γιατί η Ήτρε ψηφίζει για το ορίζον Ευρώπη και άλλα σημαντικά. Μπάζα, BASA. Είναι η συμφωνία της Βαρκελόνης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών σε ό,τι αφορά ε, την κανονιστική ρύθμιση, συγκεκριμένα συμφωνία σχετικά με τη συνεργασία για την κανονιστική ρύθμιση της ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας. Ήδη έχει τεθεί σε ισχύ αυτή η συμφωνία, η μπάσα, αλλά απαιτείται κάποια επικαιροποίηση και αυτό έγινε με την τροποποίηση που υπέγραψαν τα συμβαλόμενα μέρη στις, ε, το Δεκέμβριο του 2017 για ενίσχυση Τη εταιρική σχέση μεταξύ των δύο πλευρών. 13 Δεκεμβρίου του 2017 λοιπόν υπογράφηκε, αυτό το κείμενο για κοινού στόχου. Ε, κοινέ κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τον τομέα τη αεροπορία. Η πολιτική αεροπορία ξέρουμε ότι συνεισφέρει με πάνω από 500 δισεκατομμύρια ευρώ στο ΑΕΠΑ της Ένωσης ε, της ΥΟΣ και απασχολεί πάνω από 9 εκατομμύρια άτομα είναι ένας από τους ε, πιο αξιό, μάλλον ένας από τους ε, τομείς της οικονομίας που περισσότερο εξαρτάται από τη ρύθμιση. Ζητεί τώρα το Συμβούλιο από το Κοινοβούλιο να δώσει τη σύμφωνη γνώμη του στην έγκρισή του ε, στην τροποποίηση αυτή της συμφωνίας. Η πρόταση της Τερέσα Γκρίφιν είναι να τη δώσουμε την έγκριση αυτή για να συνεχίσει να ισχύει αυτή η πολύ ζωτική συμφωνία και να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η συνεργασία. Άρα θα δώσουμε θετική άποψη για την τροποποίηση αυτή. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ την εισηγήτρια και εσάς που την ε, αντικαταστήσατε. Και περνάμε στους σκιώδεις εισηγητέ. Για το ΕΛΚΑ θα ήθελε να πει κάτι ο Βιμ, ο Βιμ Φαντενκάμπ. Δεν ξέρω ποιος είναι σκιώδης εισηγητής εκ μέρους του ΕΛΚ για την έκθεση αυτή. Εγώ. Τέλο πάντων, λέω πρώτος, δεν βλέπω κανέναν άλλον ε, στον ε, κατάλογο. Safety first. Δεν θα έπρεπε να ισχύει μόνο για τι οδικέ αλλά και για τι αεροπορικέ μεταφορέ, κατά την άποψή μου, αυτή η αρχή πρώτη ασφάλεια. Ούτε από την Κομισιόν θέλει κάποιο το λόγο. Οπότε για τι τροπολογίε προθεσμία είναι 26 Νοεμβρίου στι 5 το απόγευμα. Σε αυτό μπορούμε να πούμε ένα ναι, ένα όχι μόνο, όπως ξέρετε αγαπητοί συνάδελφοι. Άρα μόνο αν θέλουμε να απορρίψουμε θα καταθέταμε τροπολογίες, αλλά μας συνιστά η μας να αποδεχθούμε αυτή την τροποποίηση είπα ότι ήταν το τελευταίο σημείο της σημερινής διάταξης για τη δημόσια συνεδρίαση. Περνάμε στην και κλεισμένο των θυρών συνεδρίας. Παρακαλώ όλους ε, τους ε, προσκεκλημένους να αποχωρήσουν. Ε, θα κλείσει και η μετάδοση στο διαδίκτυο. Θα παραμείνουν μόνο οι βουλευτές. Μπορείτε να τα δείτε και στην τηλεόραση, λέω, στην ομάδα επισκεπτών, γιατί μεταδιδόμαστε ζωντανά και μάλιστα με μετάφραση σε όλες τις επίσημες γλώσσες μία μικρή διακοπή και συνεχίζουμε και κλεισμένων των θυρών με την κυρία Μάισνερ.